να λαμβάνονται υπόψη και οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Ήταν κάπως ε, μονοπλευρό, το, ε, μονοβαρές ε, το παιχνίδι μέχρι τώρα. Θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει πιο ισόρροπη συμμετοχή. Νομίζω ότι είπατε αυτά που είχατε να πείτε. Επιτρέψατε μου να απαντήσω. Αυτά τα οποία κάνω, τα κάνω αναλογικά με τα αιτήματα τα οποία έλαβα για να ανταποκριθώ και στο χρόνο λειτουργίας και στην απόδοση του λόγου σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, Επίτροποι ένα ψήφισμα το οποίο έχει κατατεθεί θα ψηφιστεί αύριο στι 11.30. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη συζήτηση. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, έχουμε δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία. Κύριε Κρέιτον, σα δίνω το λόγο. Δεν είμαι βέβαιη ότι θα ενταχθεί η Τουρκία πριν από το τέλο τη Ιρλανδική Προεδρία, αλλά θα μα κάνετε εσεί μια ενδιαφέρουσα εισαγωγή για τη συζήτηση. Thank you, Madam President. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, εκ μέρου του Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη δουλειά που έχει κάνει επί του θέματο, ιδίω την εισηγήτρια κυρία Όμεν Ρόιταν. Το ψήφισμά σας τονίζει αρκετά σημαντικά θέματα και φτάνει σε μια σημαντική στιγμή στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η Τουρκία είναι και υποψήφια χώρα και βασικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τουρκική οικονομία συνεισφέρει στην ευημερία της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Η ενεργός ε, εξωτερική πολιτική της Τουρκίας σαφώς ε, έχει αυξανόμενη σημασία για όλη την περιφέρεια και ε, για τον εντυνόμενο διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Η σχέση με την Τουρκία είναι αρκετά παλιές και φαίνεται ο βαθμός στον οποίο έχουμε κοινά συμφέροντα. Ωστόσο, η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας δεν έχει επιτύχει το πλήρες δυναμικό της. Αυτό θα μπορέσει να συμβεί μόνο μέσω της πρόοδου και στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης και σε όλες τις ε, πτυχέ αυτής της σχέση. Είναι λοιπόν ενθαρρυντικό το ότι τώρα υπάρχει μια νέα δυναμική στα θέματα της ένταξη της Τουρκίας ε, με το άνοιγμα του σημαντικού ε, κεφαλαίου για την περιφερειακή πολιτική τους επόμενους μήνες και ελπίζοντας και ελπίζουμε και πριν λήξει η Ιρλανδική Προεδρία. Θα, περιμένουμε, θα περιμένω να υπάρξει ε, πρόοδο και να καταβληθεί η προσπάθεια κυρίως από τουρκική πλευρά. Ενθαρρύνουμε ε, την Τουρκία σε σχέση με αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα και από την Επιτροπή και από τους εταίρου από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση η θετική ημερήσια διάταξη θα αποτελέσει συμπλήρωμα στις διαπραγματεύσεις, δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο των διαπραγματεύσεων. Συνταγματική μεταρρύθμιση είναι το κλειδί για την πρόοδο. Στο σχέδιο ψηφίσματος τονίζεται ότι το Συμβούλιο ε, χαιρετίζει ε, το ότι η δουλειά τη Τουρκία στο νέο Σύνταγμα αποτελεί τμήμα μια ε, ευρύτερη διαδικασία δημοκρατική συνεργασία. Αυτό θα δημιουργήσει το πλαίσιο για περαιτέρω εξελίξει και για, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το κουρδικό ζήτημα. Το κουρδικό ζήτημα μας ενθαρρύνουν οι τελευταίες εξελίξεις ε, στο πλαίσιο ενευτικής ε, διαδικασίας ε, και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες θετικές πρόοδοι. Η έκκληση του Αμπτουλάου Τσαλάν προς το ΠΚΚ να καταθέσει τα όπλα είναι ενθαρρυντική, είναι μια θετική εξέλιξη θα πρέπει να συνεχίσει η πρόοδο στα συνταγματικά ζητήματα και ε, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Τουρκία θα πληρεί πλήρως τα ε, πρότυπα για την, ε, τα κριτήρια για την ένταξη. Η συνταγματική μεταρρύθμιση δεν ήταν το μόνο σημαντικό σημείο. Υπάρχει και το θέμα της δημιουργίας ενός διαμεσολαβητού και ενός θεσμικού οργάνου σε εθνικό επίπεδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει επιτευχθεί πρόοδος και για τα δικαιώματα δικαιώματα των γυναικών και για την ισότητα των φύλων με την έγκριση του τρίτου πακέτου τροποποιήσεων της νομοθεσίας και όσον αφορά τα σώματα ασφαλείας. Αναγνωρίζουμε όμως ότι απαιτείται ε, περαιτέρω προσπάθεια. Ζητούμε από την Τουρκία να συνεχίσει να τηρεί την, τα ανθρώπινα δικαιώματα και όσον αφορά την νομοθεσία και στην πράξη. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την, το δικαίωμα ελεύθερη έκφρασης. Είδαμε ότι υπάρχουν υπάρχουν πολλέ δικαστικέ υποθέσει κατά συγγραφέων και ακαδημαϊκών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι εκφράζουν τι μη βίαιε απόψει του και πολύ συχνά υπάρχουν και απαγορεύσει ιστοσελίδων. Η εφαρμογή τη νομοθεσία σχετικά με την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα παραμένει επίση μια σημαντική ε, ανησυχία και είναι θεμελιώδου σημασία να υπάρξει ανεξαρτησία και αμεροληψία για το δικαστικό τομέα, όπω και αποτελεσματικότητα. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο μέσω τη νομοθεσία, αλλά και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία. Και υπάρχουν και άλλα θέματα όπου απομένουν πολλά να γίνουν. Και εδώ ε, θα ήθελα να αναφέρω ε, την ε, ελευθερία άσκηση θρησκευτικών δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των γυναικών, των παιδιών, την καταπολέμηση τη διακριτική μεταχείριση, την καταπολέμηση των βασανιστήριων. Επίση, ένα ζήτημα που αποτελεί εμπόδιο για τι διαπραγματεύσει με την Τουρκία είναι ότι ε, η Τουρκία παρότι τις ε, επανειλημμένες εκκλήσεις μας ε, δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το συμπληρωματικό πρωτόκολλο στη Συμφωνία Ένταξης. Η θέση μας είναι απολύτως γνωστή από αυτού. Δεν υπάρχει πρόοδος στην πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλλου χωρίς διακρίσεις και όσο δεν υπάρχει πρόοδος θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζει αυτά τα οποία είχαμε πει από το 2006 και επομένως εμποδίζεται η συνολική πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Αναμένουμε από την Τουρκία να επιτύχει ε, πρόοδο και στην ε, ρύθμιση των σχέσεών της με την, ε, την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς καθυστέρηση. Ναι, είναι λυπηρό το ότι η Τουρκία πάγωσε τις σχέσεις της κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας το, το, το εξάμεινο της Κυπριακής Προεδρίας πέρυσι. Η Προεδρία είναι ένα βασικό τμήμα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να χαίρει αντίστοιχου σεβασμού. Επίσης θα ήθελα να τονίσω τη σημασία την οποία γενικά αποδίδουμε στις, κανέ, στις καλές ε, σχέσεις γειτονίας. Είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την μέτρηση της προόδου της Τουρκίας προς ε, την ε, οδό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κλείνοντα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό θέμα των διμερών σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία, δηλαδή την απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίου. Υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου που ζητεί από την Τουρκία να λάβει βήματα προ την απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίου ω ε, μια μακροπρόθεσμη προοπτική παράλληλα με την ε, υπογραφή τη συμφωνία Επανεισδοχή. Το Συμβούλιο ε, υποστηρίζει το διάλογο για τι θεωρήσει διαβατηρίου και για τη μετανάστευση και ταυτόχρονα είναι θεμελιώδου σημασία ε, η συμφωνία επανεισδοχή που έχουμε διαπραγματευτεί με την Τουρκία να υπογραφεί και να ε, συναυθεί και να τηρείται στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και δίνω το λόγο στον κύριο Φιούλε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, αξιότιμα μέλη, θα ξεκινήσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια, την κυρία Μενράιτεν πολύ μεγάλη ποιότητα της εκθέσεως που συζητούμε σήμερα. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρωπα... σε σχέση Ευρωπαϊκής Ενώσεως Τουρκίας ε, δημιουργούν αίτια αισιοδοξία. Στο Συμβούλιο του περασμένου Δεκεμβρίου αναφέρθηκε νέα ορμή και προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να αρχίσουμε κεφάλαια των διαπραγματεύσεων ξανά το 2013. Δεύτερον, Σημειώνουμε πρόοδο στην συνεργασία μα όσον αφορά τη μετανάστευση και τι θεωρήσει. Όπω αναφέρθηκε μόλι τώρα, έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε σύντομα να αρχίσουμε ένα διάλογο για τι θεωρήσει με την Τουρκία μαζί με την υπογραφή τη Συμφωνία Επανεισδοχή με την Τουρκία και, μεταξύ Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δύο εβδομάδε πριν από δύο εβδομάδε, το Τουρκικό Κοινοβούλιο θέτησε το νόμο για του αλλοδαπού και τη διεθνή προστασία. Από τη στιγμή θα εφαρμοστεί αυτό σωστά, αυτό ο νόμο θα καλύπτει και κάποια σημαντικά ζητήματα ε, περί του δικού χάρτου για τις θεωρήσεις τρίτων. Διάλογος για την εξωτερική πολιτική μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει εντατικοποιηθεί. Ε, ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένη ευθυγράμμιση της Τουρκίας με τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εκτιμούμε και υποστηρίζουμε τη συνεχή ενεργό ε, δράση της Τουρκίας για τη Συρία και τον ζωτικό ρόλο της, τον ανθρωπιστικό και την αντιμετώπιση της εισρωής των Σύρων προσφύγων. Πάνω από 190.000 καταγεγραμμένους ε, πρόσφυγες ε, φιλοξενεί η Τουρκία. Η προσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι κάτι καλό και αυτό αξιότιμα μέλη θα, αρχίσει θα υπογραμμίσω και πρόσφατες εξελίξεις εντός της χώρας. Η σύνταξη ενός ε, καινούριου συντάγματος έγινε μια, σε μια κρίσιμη καμπή. Η, η συμμετοχική διαδικασία ακολούθησε σωστό δρόμο και την υποστηρίζουμε πλήρως νέα πρωτοβουλία για ειρήνη επιτέλους στα νοτιοανατολικά της χώρας ε, είναι μια ευκαιρία που υπόσχεται το τέλος της τρομοκρατίας και ανοίγει το δρόμο για γενική λύση του κουρδικού προβλήματος. Το τέταρτο πακέτο μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου που θετήθηκε από το τουρκικό κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα είναι σημαντική εξέλιξη όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Δεν εξαιρεί την κυβέρνηση από την θέσπιση κι άλλων μεταρρυθμίσεων. Παραμένουν διατάξεις στην τουρκική νομοθεσία που δημιουργούν ανησυχίες. Κυρίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία ε, του, της ενελεύσεως ε, και της ε, ομαδικής συμμετοχής. Ε, τα εκκρεμή σημεία από ό,τι κατάλαβα θα συμπεριληφθούν στη, στο επικείμενο σχέδιο δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Όσον αφορά το κυπριακό ζήτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει σε επανέναρξη πλήρων διαπραγματεύσεων το ταχύτερων δυνατόν με στόχο την επίτευξη ταχείας ε, ολοκλήρωσης των συνομιλιών παρόλο που κατανοούμε ότι άμεση προτεραιότητα της δημοκρατίας της Κύπρου ε, είναι αλλού. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ταμπού στην προσπάθεια για μια γενική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος. Ελπίζω ότι το γενικό θετικό κλίμα που προανέφερα στην αρχή της παρέμβασής μου θα μεταμορφωθεί σε ευκαιρία και δυνατότητα που θα είναι προς και της ελληνοκυπριακής κοινότητας και της τουρκοκυπριακής. Μια διευθέτηση θα συμβάλλει σημαντικά σε καλύτερο επιχειρηματικό, διαμόρφωση καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και θα απελευθερωθεί το πλήρες οικονομικό δυναμικό του νησιού και στον τομέα τον ενεργειακό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Όμεν Ρόιτεν για αυτό. Ναι. Κυρία Όμεν Ρόιτεν, έχει τον λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Ποτέ δεν ήταν βαρετή η ατμόσφαιρα όταν γίνεται λόγος για τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Πολλά τεκταίνονται πρόσφατα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την τέταρτη αναθεώρηση σε σχέση με τα θέματα δικαιοσύνης που υιοθετήθηκε από την Τουρκική Βουλή και θα συμφωνούσα με ε, την Επιτροπή και την κυρία Κράιτον ότι πρέπει να συμπληρωθούν σε σχέση με τις προθέσεις αυτές οι διαβουλεύσεις και αυτός ο διάλογος. Μετά έχουμε και το πρόγραμμα δράσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου που φαίνεται ότι καταλήγει και αυτό σε το πρόγραμμα σε κάποιες πιο θετικές εξελίξεις. Έχουμε επίσης ε, και τον νόμο, το νομοθέτημα περί αλλοδαπών εδώ και αρκετό χρόνο υπό εξέταση. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν με την κυβέρνηση και τον κύριο Οτζαλάν φαίνεται ότι συνεχίζονται επικοδομητικά με μεγάλη υποστήριξη των Τούρκων πολιτών. Αυτό είναι εκείνο το οποίο εκτιμούμε ιδιαίτερα. Την υποστήριξη των ίδιων των Τούρκων πολιτών για αυτή τη διεργασία και την υποστήριξη των μελών της κοινωνίας των πολιτών εξίσου. Επίσης και μια βελτίωση φαίνεται να αναφύεται σε σχέση με τις ε, σχέσεις ε, Τουρκίας και Ισραήλ σε σχέση με τα πρόσφατα συμβάντα. Επίσης ε, και η γαλλική κυβέρνηση απέσυρε απαγόρευση ε, όσον αφορά το κεφάλαιο 22, όσον αφορά την Τουρκία και ελπίζουμε ότι θα σημειωθεί πρόοδο στου επόμενου μήνε. Αναφέρθηκε σε σχέση με το κεφάλαιο 19 κοινωνική πολιτική που θέλουν να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο και να εξεταστεί. Δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέχρι σήμερα. Φαίνεται ότι άλλαξαν άποψη και αυτό είναι θετικό. Αυτό είναι το γενικότερο σκηνικό εν ώψη του οποίου συζητούμε αυτό το ψήφισμα σήμερα. Ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω επικοδομητική σχέση με την Τουρκία. Επικοδομητική μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων φυσικά. Αλλά για να επιτευχθεί αυτό ο στόχος, αμφωτέρωθεν χρειαζόμαστε μια δέσμευση, στεναρή βούληση από την Τουρκία και σε σχέση με το 2005 ήδη Υπάρχει ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, όχι επειδή επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλυθούν μεταρρυθμίσεις από την Τουρκία, αλλά προς όφελος της ίδιας της Τουρκίας. Αν οι Τούρκοι θέλουν να είναι ένα σύγχρονο κράτος, μια σύγχρονη κοινωνία, πρέπει να συνεχίσουν τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και φυσικά είναι εξίσου σημαντικό η ελευθερία της έκφρασης. Όλα αυτά. Έχω τρία λεπτά, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε. Λοιπόν, και οι βασικές θεμελιώδεις ελευθερίες όπως ε, τα δικαιώματα των θρησκευτικών κοινοτήτων ε, κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι η Τουρκία βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε και το θέμα όλα της ε, βούλησης και της ίδιας της νοοτροπίας στην προσέγγιση αυτών των θεμάτων. Αν δούμε τις, τους τριμερείς διαλόγους υπάρχουν φυσικά σε κάποια θέματα κάποια προβλήματα. Υπάρχει εδώ ένα ε, ισόρροπο ε, ψήφισμα και ε, καλοχαιρετίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, ασκούνται όμως επικρίσεις εκεί όπου είναι αναγκαίο. Θα θέλαμε να πούμε ότι έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα, αν δραχθούμε αυτή τη ευκαιρία, η Τουρκία με μια νέα κυβέρνηση στην εξουσία, με μια νέα κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, να αντιμετωπίσει το κουρδικό πρόβλημα με αποφασιστικό, με στεναρό τρόπο. Με συμφωνίε με του Κούρδου που ελπίζουμε ότι θα σημειωθούν φέτο. Ευχαριστώ. Αν δούμε την κατάσταση τόσο και στην Τουρκία όπως και στην ευρύτερη περιοχή καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια μεγαλύτερη προσπάθεια για τις επικοδομητικές σχέσεις ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία είναι απόλυτα αναγκαίο στοιχείο αυτές, αυτή η επικοδομητική σχέση. Αυτός είναι ο εστιασμός, η επικέντρωση της έκθεσης. Μια έκθεση συνενετική ουσιαστικά και που θα τύχει μεγάλης πλειοψηφίας όπως ελπίζουμε σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και σε αυτή τη διαδικασία εκπόνησης έκθεσης από πλευράς της εισηγήτριας δράτω με τις ευκαιρίες να συγχαρώ την κυρία Ομερόιτεν Ρόιτεν ως εισηγήτρια η ομάδα μας ουσιαστικά είχε τρεις προτεραιότητες η πρώτη από αυτές τις προτεραιότητες ήταν να ενισχύσει τις θετικές και γόνιμες σχέσεις με την Τουρκία η ανάπτυξη αυτή της ε, θετική πτυχή σε διάφορες πτυχέ, η αναζήτηση θέσεων από την άλλη πλευρά που θα είναι το δυνατόν ευρύτερα κοινέ και θα τι συμμεριζόμαστε στον μέγιστο βαθμό με την Τουρκία σε σχέση με μια περιοχή δηλαδή στη Μέση Ανατολή που έχει ιδιαίτερα προβλήματα που ε, αντιμετωπίζει. Και η δεύτερη προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε και να σημειώσουμε πρόοδο, να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός στι διαπραγματεύσεις ε, για την ένταξη, με, την, με το άνοιγμα νέων κεφαλαίων. Και η τρίτη προτεραιότητα, χωρίς να αναμειχθούμε με κανένα τρόπο στα εσωτερικά της Τουρκίας, είναι η αναζήτηση υποστήριξης για την, τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Συμβαίνουν εκεί πολύ σημαντικά πράγματα. Αφενός η ανάπτυξη μια σειρά μεταρρυθμίσεων όσον αφορά την νομοθεσία, για το δικαστικό σώμα, για τα, το, το δικαστικό σκέλος, τα δικαιώματα των γυναικών. Υπάρχουν εδώ και ε, θέσεις ε, που είναι ίσως αντιφατικές. Πρέπει όμως να υποστηρίξουμε τις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε όλους αυτούς τους τομείς. Υπάρχει και μια διαδικασία συνταγματική που έχει τεράστια σημασία. Και τέλος υπάρχει και μια διαδικασία ειρήνευσης, ειρηνικής συμβίωσης. Μετά από δεκαετίες σειράξεων που στήχησαν μυριάδες θύματα και δισεκατομμύρια δολάρια σε χρήματα, τώρα υπάρχει μια ευκαιρία συμφιλίωση Τούρκων και Κούρδων και πρέπει εδώ να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δώσει ενεργά τη συνδρομή τη. Ευχαριστώ κύριο Λάμστοφ τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και φέτος το Ευρωκοινοβούλιο αποστέλει ένα μήνυμα προς την Τουρκία που έχει δύο μέρη Αφενό υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων, δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία. Από την άλλη πλευρά έτοιμα για περισσότερε μεταρρυθμίσει και ταχύτερη πρόοδο. Είναι τώρα η χρονική στιγμή αναμφίσιμα να δείξει η Τουρκία ότι ενδιαφέρεται για περαιτέρω μεταρρυθμίσει σε ευρύτερο πλαίσιο. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι εσεί, Επίτροπε και εσεί, Υπουργέ, λέτε ότι υπάρχουν κάποιε πρόοδοι στο διαμεσολαβητή, σε κάποια άλλα θέματα. Όμω μετά από αυτά τίθενται σημαντικά ε, ζητήματα, θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθερία της έκφρασης, πολιτικά δικαιώματα. Είναι αποφασιστική σημασία. Η Άγκυρα πρέπει να πάρει αυτό το μήνυμα και να το αφουγκραστεί, να εισακούσει αυτό το μήνυμα. Μπορώ να επαναλάβω ότι για μια χώρα που διαπραγματεύεται για την ένταξή της ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι μια χώρα όπου οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν ελεύθερα και διώκονται και είναι η μεγαλύτερη φυλακή δημοσιογράφων παγκόσμια με η Τουρκία. Ελπίζω ότι με το τέταρτο πακέτο μεταρρύθμισης τη δικαιοσύνη, του τομέα ε, του δικαστικού και της δικαιοσύνη ε, θα γίνουν θετικά βήματα. Υπάρχουν σφάλματα και λάθο αποφάσεις που ελήφθησαν. Πρέπει να υπάρξουν μηνύματα ότι δεν θα ανεχθούμε τέτοιου είδου ε, παρεκκλήσει. Εκφράζω τη θλίψη μου ότι δεν καταφέραμε στην συνταγματική διαδικασία όσον αφορά το Συμβούλιο τη Ευρώπη και τη διαδικασία τη Βενετία να εμπλέξουμε περισσότερο πιο στενά αυτή τη διαδικασία σε σχέση με με την Τουρκία. Δεν είναι ξένη εξουσία το Συμβούλιο της Ευρώπης που αναμειγνύεται στα θέματα της Τουρκίας. Είναι ένα θεσμικό ε, όργανο στην Ευρώπη που δίνει αγώνα για τα θεσμικά και δημοκρατικά δικαιώματα και δεν μπορεί αυτό να αποκλειστεί σε σχέση με την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ευκαιρία. Η ευκαιρία που ε, διαγράφεται, αυτά από τα οποία συμβαίνουν σε σχέση με την Τουρκία, οι τοποθετήσει, οι δηλώσει του Αμπτουλά Ετζαλάν, ο θετικό ρόλο του Μπεντεπέ, του κουρδικού αυτού κόμματο, είναι ένα σταυροδρόμι, μια σημαντική ιστορική ευκαιρία. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουν οι Τούρκοι το θέμα τη υπηκότητα, τη ηθαγένεια, ε, των νομοθετημάτων κατά τη τρομοκρατία ε, να τα ρυθμίσουν οι Τούρκοι με τέτοιο τρόπο εξάπαντο και να υπάρξει ειρήνη σε σχέση με του Κούρδου και την Τουρκία. Αυτό αξίζει και πρέπει να γίνει. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Τουρκία βρίσκεται σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Τώρα πρέπει αξιόπιστα η Τουρκία να προαγάγει τι μεταρρυθμίσει και να συνεχίσει αξιόπιστα την ευρωπαϊκή πορεία τη υλοποιώντα ε, τι προποθέσει που έχουν τεθεί ώστε να σημειωθεί πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάνστροφ. Κυρία Φλότχ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι αλήθεια ότι στο Κοινοβούλιο δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να καταρτίζουμε μια έκθεση σε μια χρονική στιγμή τόσο σημαντική όσο είναι αυτή, τη στιγμή, αυτή η χρονική στιγμή για την Τουρκία και για ολόκληρη την περιφέρεια και για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να συγχαρούμε την Ρία Όμεν Ρόιτεν που κατάφερε να τα βγάλει πέρα και να ετοιμάσει αυτή την έκθεση που είναι μια έκθεση πολιτικών εταίρων χωρίς να θέλει να είναι ε, ε, κυδεμονευτική και αντιμετωπίζοντας θέματα θέματα που έχουν μεγάλη πολιτική ευαισθησία, όπω είναι το δικαίωμα των μειονοτήτων, η ελευθερία έκφραση, η κατάσταση των γυναικών, τα αναφέραμε μόλι, ή τα θέματα του περιβάλλοντο και νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ χρήσιμη στην τωρινή κατάσταση που είναι μια ιδιαίτερα σημαντική κατάσταση διότι ε, και στις διπλωματικές σχέσεις ε, και στις, ε, στα πολιτικά πράγματα γίνονται σημαντικές αλλαγές. Η πολιτική αλλαγή στην Γαλλία έχει δημιουργήσει νέες καταστάσεις. Το βέβαιο για το κεφάλαιο 22 είναι κάτι το οποίο δημιουργεί νέες συζητήσεις και ε, η ειρηνευτική διαδικασία που ξεκινάει από την ε, τουρκική κυβέρνηση με ε, τους Κούρδους είναι μια σημαντική διαδικασία και είναι κρίμα που χρειάζονται πάνω από 40 μέλη για, ε, σχετικά ε, με τα κεφάλαια 23-24, διότι όποιος θέλει να μιλά για, τα, ε, για την κατάσταση στην Τουρκία θα πρέπει να μπορεί και να υποστηρίξει τη σημαντική δύναμη που κρύβεται πίσω από αυτά τα δύο κεφάλαια που αφορά θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, θέματα δικαιοσύνης και του δικαστικού σώματος. Η τροπολογία αυτή λοιπόν είναι πραγματικά ε, λυπηρή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα στην Τουρκία, όπως σας έλεγα, συμβαίνουν πράγματα που δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει πλήρως την ευρύτητά τους. Ε, ε, υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ του κυρίου Τσελάν που είναι στη φυλακή και του κυρίου Ερντογάν που έχει μεγάλη υποστήριξη από την κοινωνία των πολιτών και αυτό είναι πολύ σημαντικό και συνδέεται και με τη συζήτηση για το νέο σύνταγμα. Εφόσον το θέμα του ορισμού της ηθαγένειας, το θέμα της δυνατότητας εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα, το θέμα της αποκέντρωσης και του εκδημοκρατισμού στην Τουρκία συνδέεται με την ε, πολιτική επίλυση του θέματος των Κούρδων και της ειρηνευτικής αυτής διαδικασίας. Νομίζω λοιπόν ότι η έκκληση όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προς την κατεύθυνση αυτή έχει κέρια σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να προσφέρει. Την εμπειρία της καταρχήν στα θέματα ειρηνευτικής διαδικασίας, την ικανότητά της να δημιουργήσει πολιτικού συμβιβασμού, πολιτικό διάλογο και σεβασμό στον πολιτικό διάλογο γιατί είναι κάτι το οποίο λείπει ακόμη καταφανώς στην τουρκική πολιτική ζωή. Έχετε μια μπλε κάρτα, τη δέχεστε? Μάλιστα, μάλιστα. Ο κύριος Ντάρμουθ. Κυρία Πρόεδρε, βλέπω ότι έχετε εκλεγεί ως πράσινη και μιλώντας για την Τουρκία, διερωτώ με, κάνατε μια αξιολόγηση Ποια είναι η συνέπεια στο περιβάλλον για τη χώρα σας. Δηλαδή σε 73 εκατομμύρια Τούρκους πολίτες να δώσετε το απόλυτο δικαίωμα να εργαστούν, να ζήσουν και να εγκατασταθούν στη Γαλλία. Το σκεφτήκατε αυτό. Ε, κυρία Φλότρο, ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξέρετε ότι οι τροπολογίες που αφορούν ακριβώς τις ανησυχίες που έχουμε όσον αφορά τον τρόπο ανάπτυξης αρκετά που υποστηρίζει πολύ την παραγωγή και την ανάπτυξη του παλιού μοντέλου στην Τουρκία, αυτά εκφράστηκα από την ομάδα μου και είναι στην έκθεση της κυρίας Όμεν Ρέιτεν. Κατά τα λοιπά δεν ξέρω πολύ καλά τι θέλετε να πείτε όσον αφορά την περιβαλλοντική συνέπεια της προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα είμαι στην πρώτη γραμμή για αυτά τα θέματα, στη συζητήση με τους ομολόγους μας στην Τουρκία για, για την αλλαγή του κλίματος, ε, για την καταπολέμηση κατασκευής πυρηνικών αντιδραστήρων στην Τουρκία, για να φροντίσουμε ούτως ώστε η ανάπτυξη της Τουρκίας να είναι πλούσια σε απασχόληση αλλά και πλούσια σε κοινά αγαθά όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κύριε Φλότρο και Τώρα πάμε στη σειρά την κανονική που το λόγο τον έχει ο κύριος Τάνο και δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι οικονομικός και πολιτικός κινητήρας η Τουρκία για την Ασία και την Ευρώπη και είναι και στις δύο επίρους. Ε, και πάντα είχε θέση στην ιστορία και λόγω γεωπολιτικών και κοινωνικών πραγματικότητων σήμερα. Και η ECR παραδέχεται ότι η Τουρκία είναι σημαντική και προσπαθεί να ενισχύσει του δεσμού μα και τη συνεργασία με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια δημοκρατία που επιθυμεί στενότερη ολοκλήρωση ευρωπαϊκή ενώ οικοδομή και σχέση στη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία. Πράγματι, κάποιε αυτέ οι σχέσει θα πρέπει να είναι άκρο επρόσδεκτε από το Κοινοβούλιο. Η προσέγγιση με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ καλά μαντάτα για εκείνου από εμά που υποστηρίζουν πιο σταθερή Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο. Και οι δύο πλευρέ θα πρέπει να τύχουν συγχαρητηρίων για τι προσπάθειε που καταβάλουν. Επίση, είναι τεράστια ενθάρρυνση που ακούσαμε πρόσφατα ότι έγινε κατάπαυση του πυρό από πλευρά του ΠΚΚ και άρχισε διάλογο με τον Σαλάν που στη φυλακή. Παρ' όλα αυτά, απομένουν προκλήσει για την Τουρκία και για τη σχέση Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί από εμά είμαστε άκρω απογοητευμένοι συγκεκριμένη, διότι αρνήθηκε να συνεργαστεί η Τουρκία με τη Δημοκρατία τη Κύπρου κατά τη διάρκεια τη Προεδρία του Συμβουλίου ε, πέρσι. Και θα είναι πολύ δύσκολο να εξετάσουμε τον ενδεχόμενο προσχώρηση τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το θέμα τη αναγνώριση τη Κύπρου παραμένει εκρεμέ. Και η Τουρκία επιμένει μονομερό να αναγνωρίζει την, το TRNC, τη Δημοκρατία τη Βορειάς Κύπρου, ε, όπως αποκαλείται, και δεν επικυρώνει το πρωτόκολλο ε, της, ε, που έχει υπογραφεί και με τους αλαφίτες στη Συρία ε, ε, πρέπει να δούμε θα γίνει και υποστηρίζει την, τον ελεύθερο στρατό της Συρίας που, κατα, πολεμά το καθεστώς του Ασάντ. Ε, αλλά υπάρχει κίνδυνος να αποσταθεροποιηθεί περαιτέρω η περιοχή και η Τουρκία. Θα, πρέπει να υποστηρίξει περισσότερο τις μειονότητες στην Τουρκία. Είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι Σύριοι, ή ε, επίση και ομοφιλόφιλοι και λοιποί θα πρέπει να ληφθούν σοβαρότερα υπόψη. Παρά όλα αυτά τα προβλήματα και τι προκλήσει, επαναλαμβάνω ότι από την έποψη του ECR η Τουρκία εξακολουθεί να είναι βασικό φίλο και σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να τίνουμε χείρα διαλόγου και συνεργασία προ την Τουρκία και να βοηθήσουμε το λαό τη και την κυβέρνησή τη να πετύχουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που επιδιώκουν διακαώ. Ε. Σα ευχαριστώ, συνάδελφε Τάνο. Τώρα θα λάβει λόγο για 1,5 λεπτό ο κύριο Μπέλντερ εξ ονόματος της Ευρώπης των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αύριο έξι χρόνια συμπληρώνονται από τότε που η τριπλή ας την αποκαλέσουμε έτσι πρωτοβουλία. Ε, η τριπλή αυτή εκδήλωση σε σχέση με τα θύματα την προηγούμενη εβδομάδα εξεφράστη η ελπίδα ότι σε σχέση με τα όσα συνέβησαν με τον σύζυγό της θα υπάρξει αποκατάσταση. Υπάρχει αυτό το τρομερό ερώτημα, Επίτροπε σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Υπάρχει κάποια ελπίδα. Η δίκη ακολουθεί βραδύτα τους ρυθμούς. Υπάρχει κάποια ελπίδα να υπάρξει διαφάνεια. Η Τουρκία θέλει να είναι ένα κράτος δικαίου και οι μειονότητες οι θρησκευτικές όπως οι χριστιανοί θα έπρεπε να αξίζουν να τύχουν υποστήριξης. Τι γίνεται λοιπόν σε σχέση με αυτή τη δίκη. Και μία άλλη ερώτηση, πάλι σε σχέση με, αυτό το, με αυτή τη δίκη, πάλι την προηγούμενη εβδομάδα αφορά αυτό ο συνήγορος των ε, οικογενειών των θυμάτων απειλήθηκε με δολοφονία. Απείλησαν να τον δολοφονήσουν. Οι ε, τουρκικές αρχές κάνουν αυτό το οποίο είναι αναγκαίο για να προστατευτεί η προσωπικότητα αυτού του δικηγόρου, να προστατευτεί ο δικηγόρος αυτός θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση στις ε, τουρκικές αρχές ε, να αναλάβουν δραστήρια ε, αποτελεσματική δράση να αντιμετωπιστούν αυτά τα συμβάντα. Και το ίδιο ισχύει και για την εβραϊκή κοινότητα. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να ενθαρρύνουν την Τουρκία να παράσχει υποστήριξη και συνδρομή. Για παράδειγμα σε σχέση με Εβραίου ε, εκδότε που απειλούνται στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Μπέλτερ. Από πλευρά Ενωτική Αριστερά θα λάβει τώρα τον λόγο για 1,5 λεπτό κύριο Χαζηγεωργίου παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι μερικά χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο και έχω την εντύπωση ότι αυτή η έκθεση ουσιαστικά σιγά σιγά αντικατοπτρίζει τις ισορροπίες μέσα στο Κοινοβούλιο αντί να κοιτάξει τα βαθιά δομικά προβλήματα της Τουρκίας. Αυτό δεν πρέπει να είναι δουλειά των Ευρωβουλευτών. Μπορεί να είναι δουλειά των κυβερνήσεων, να είναι δουλειά των διπλωματών, μπορεί να είναι δουλειά των, ε, ε, της Επιτροπής. Δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να δουλεύει με έναν τρόπο που να κρατά τις ισορροπίες μη θυμώσει ο α ή ο β. Το κουρδικό ζήτημα είναι, είναι ένα τεράστιο θέμα. Πώ έσπρωξε ποτέ αυτή η έκθεση προ τη σωστή κατεύθυνση. Εδώ οι άνθρωποι έβαλαν στη φυλακή κάποιον διότι στην προθήκη του καταστήματο του είχε μια φωτογραφία και η φωτογραφία έμοιαζε του Οτσαλάν. Και μου λένε ότι κάνουν διαπραγματεύσει με τον Οτσαλάν. Υπάρχει μια κοροϊδία. Ε, η Τουρκία δεν είναι έτοιμη να κινηθεί προ τη σωστή κατεύθυνση επίλυση ενό παραδέχομαι πολύ μεγάλου και τεράστιου προβλήματο. αλλά εμεί, αν θέλουμε να βοηθήσουμε πρέπει να είμαστε ειλικρινεί, να δώσουμε κατευθύνσει. Ε, τις λύσεις και όχι απλώς ε, κουβέντες. Όσον αφορά το Κυπριακό, κάθε χρόνο η έκθεση λέει να αποσυρθούν άμεσα τα τουρκικά στρατεύματα και να παραδοθεί η πόλη της του ε, στους κατοίκους της. Τι απαντά πίσω η Τουρκία. Υπάρχει λέει ανισορροπία μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή μας κοροϊδεύει στο τέλος ότι έχουμε μια ανισορροπία μέσα στο κεφάλι μας. Αυτή είναι η αντιμετώπιση της Τουρκίας. Οι απειλές της ενάντια στα δικαιώματα της Κύπρου να ε, εκμεταλλευτεί τον, τον υποθαλάσσιο πλούτο της. Δίνει αυτό ευκαιρία στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος να επιτρέψει να ανοιχθεί το κεφάλαιο της ενέργειας όπως απαιτεί η έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Τάκη. Ο κύριος Νταφ τώρα παρακαλώ. Εσείς έχετε σημειωθεί εδώ για να παρέμβετε για αυτό το θέμα, εντάξει θα κάνετε την ερώτηση. Αν κάνετε την ερώτηση μετά δεν θα παρέμβετε ω αγορητή στη συνέχεια. Εσείς να επιλέξετε. Θέλετε τώρα να υποβάλλετε ερώτηση ή θέλετε ύστερα να παρέμβετε ω αγορητή. Αν κάνετε τώρα ερώτηση δεν θα λάβετε τον λόγο ως αγορητή στη συνέχεια από τον κατάλογο. Εσείς θα επιλέξετε τι επιθυμείτε, τι προτιμάτε καλύτερα. Πρόεδρε. Ε, δεν το είχα αξιολογήσει ότι αν ζητά κανείς να θέσει μια ερώτηση με μπλε κάρτα έτσι απεμπολεί το δικαίωμα να παρέμβει από τον κατάλογο αγορητών στη συνέχεια. Νομίζω είναι κάτι το οποίο αγνώ αυτό ως κανονισμός, ε, ως διάταξη. Κύριε Νταφ, για να επιτρέψουμε σε όλους τους συναδέλφους να παρέμβουν γίνεται αυτό, εντάξει. Κύριε Περδόν, Προσέξτε, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Σε παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Για, για δικαστικό εσείς. Ε, κύριε πρόεδρε, με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό. Παρέστηνε επανειλημμένα σε αυτέ τι συζητήσει. Είχα το προνόμιο να υποβάλω ερωτήσει με γαλάζια κάρτα, με τη σύμφωνη γνώμη του συναδέλφου επανειλημμένα. Και εσείς, κύριε μου, είστε ο μόνο πρόεδρο που έχει θεσπίσει από τον κανόνα ότι αν κάποιο μιλά σε μία συζήτηση δεν μπορεί να σηκώσει γαλάζια κάρτα. Έχετε δικαίωμα να κάνετε δικό σα τέτοιο κανόνα, σύμφωνα με το εσωτερικό κανονισμό, αλλά είναι προσωπική απόφαση και καταστέλει τη συζήτηση. Με κάθε σεβασμό σα ζητώ, κύριε μου, να το επανεξετάσετε. Λοιπόν, τα επανεξετάζω όλα. Όλα τα επανεξετάζω. Ευχαρίστω. Αλλά προσέξτε, Όλα τα επανεξετάζω πάντα, εντάξει, αλλά ολοκληρώνω πάντα τις συζητήσεις μου έγκαιρα χρονικά, στο χρόνο που προβλέπετε και παρεμβαίνουν όλοι όσοι εγγράφονται, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Τώρα, ζητάτε μία μπλε κάρτα, μία ερώτηση, δεν είναι διαδικαστικό. Διαδικαστικό αναφέρεται. Point of order. I can understand... διαδικαστικό. Καταλαβαίνω κύριε Πρόεδρε ότι μπορεί να μην θέλετε να δώσετε στον κύριο Νταφ το δικαίωμα να μιλήσει στο τέλος αλλά αν ήδη είναι στον κατάλογο αγορητών από την πολιτική του ομάδα, δεν μπορείτε να του το αρνηθείτε αυτό επειδή ζήτησε μπλε κάρτα. Μπορείτε να το κάνετε αν θέλει να παρέμβει στην διαδικασία Catch the αλλά δεν μπορείτε να τον βγάλετε από τον κατάλογο των αγορητών τη ομάδα του αν ζητήσει μπλε κάρτα. Διαφορετικά καταστρέφεται η δυναμική μια. Πολύ καλά, πολύ καλά, δόκτωρα. Τάνοκ. Ε, σημειώνω αυτή την ερμηνεία σα και σέβομαι την ερμηνεία σα. Αλλά αυτό που προεδρεύει σε αυτή τη συνεδρία σε την Ολομέλεια είμαι εγώ και θα διατηρήσω αυτή την απόφαση. Όταν θα παρέμβετε στη συνέχεια μπορείτε να σχολιάσετε ό,τι επιθυμείτε κύριε Νταφ για το θέμα αυτό που είναι υποσυζήτηση. Αναλώσαμε πολύ χρόνο. Θα λάβει τον λόγο ο κύριο Στάσεν. Εξ ονόματο των μη εγγεγραμμένων. Για 1,5 λεπτό κύριο Στάσεν. Κυρία Στάσεν παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για 1,5 λεπτό. Στο άρθρο 49 για τη Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναφέρεται ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα η οποία εφαρμόζει και σέβεται τις αρχέ μπορεί να υποβάλει αίτηση για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι όμως ευρωπαϊκή χώρα η Τουρκία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επιπλέον διαρκώς το παραβιάζει αυτέ τι αρχέ η Τουρκία. Κάνουμε λόγο για τι αρχέ και αξίε τη ελευθερία, τη ισότητας. Δεν υπάρχουν και δεν είναι σεβαστές αυτέ οι αρχέ και αξίε στην Τουρκία. Θα ήθελα απλά και μόνο να αναφέρω ότι εντάξει, πολύ ωραία να γίνει μια, ένα σύγχρονο κράτο η Τουρκία. Όμως ε, δεν ε, απομένουν πολλά. Εδώ υπάρχουν ε, ποινές ε, ε, δεκάμινες ε, και επιβολές κυρώσεων. Γιατί όλα αυτά επειδή κάποιο κείμενο από τον 10ο αιώνα του ποιητή Ομάρ Χαγιάμ θεωρείται λέει προσβολή στο Ισλάμ, εις βάρος του Ισλάμ. Απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ασκήσει την επιρροή της, να επιμείνει και να εμείνει ότι θα υπάρξουν σημαντικές συνέπειες λόγω της ποινή που επευλήθησε σε αυτόν τον πιανίστα τον Φαζίλ Σάι δηλαδή. Και θέλω πραγματικά να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή τη χώρα που δεν είναι ευρωπαϊκή, δεν θέλει να είναι ευρωπαϊκή και θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, εντάξει. Λοιπόν, τι θα κάνετε σε σχέση με όλα αυτά. Θα παραμείνετε στι θέσει σα και στι αρχέ σα και θα σταματήσουν οι διαπραγματεύσει με την Τουρκία επιτέλου ή όχι. Πρόεδρο, προσέξτε, στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Τάνοκ πιο πριν, είπα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Στάσεν. Είναι η κυρία Στάσεν φυσικά και ζητώ συγγνώμη για το σφάλμα που έκανα και άλλαξα φίλο στην κυρία Στάσεν. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο αγορητών εξ ονόματος των ομάδων και περνάμε στους αγορητές που θα παρέμβουν ατομικά. Και πρώτα απ' όλα θα το κάνει ο συνάδελφος Έλμα Μπροκ που θα παρέμβει. Δύο λεπτά για την παρέμβασή σας κύριε Μπροκ. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές. Η Τουρκία χωρίς καμιά αμφιβολία είναι ένας σημαντικός θεμελιώδους σημασίας εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταίρος που έχουμε αμοιβαία στρατηγικά συμφέροντα με αυτόν εμείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι εξελίξεις σε σχέση με την Τουρκία που καθιστούν σαφές ότι η Τουρκία στη, στο, βρίσκεται στο διατλαντικό και ευρωπαϊκό στρατόπεδο και στην ευρωπαϊκή πτέρυγα και πλευρά. Ας δει κανεί το χάρτη να καταλάβει ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης και προς το συμφέρον της Τουρκίας να αποτελεί μέρος μιας τέτοιας εξέλιξης και θα ανήκει σε αυτό το πλαίσιο και μάλιστα και με επιτυχή τρόπο να στεφτεί με επιτυχή αυτό το εγχείρημα. Βρίσκω ότι η Τουρκία είναι ένας παράγοντας σταθερότητας, μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιφέρεια, ευρύτερη περιοχή και γι' αυτό χαίρομαι για το ότι οι σχέσει μεταξύ Τουρκία και Ισραήλ έχουν βελτιωθεί και παίρνουν μια θετικότερη τροπή. Πρέπει να ενθαρρύνουμε να συνεχιστεί αυτή η πορεία ώστε να υπάρξει σταθερότητα, να σταθεροποιηθεί η περιφέρεια αυτή. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι τομεί όπου υπάρχουν ε, κάποια θέματα όσον αφορά την μεταφορά ενεργειακών προϊόντων. Και για την Τουρκία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Και ίσω θα πρέπει σε αυτού του τομεί να εστιαστούμε στι διαπραγματεύσει με αντίστοιχα πακέτα τα οποία θα εξετάσουμε ανεξάρτητα ανεξάρτητα αν θα γίνει στο τέλος τέλος κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία ή όχι, πρέπει αυτά τα θέματα να ρυθμιστούν ούτως ή άλλως. Και πιστεύω εξάλλου ότι στην έκθεση αυτή σε σχέση με την Τουρκία γίνεται λόγος για πρόοδου σε σχέση με το νομικό σύστημα, την ε, ε, ε, ελευθερία του εκφράζεσαι, θρησκευτικέ ελευθερίε, αλλά επίση καθίσταται σαφέ ότι δεν έχει πετύχει η μεγάλη αλλαγή, η μεγάλη καμπή. Και αυτό είναι το αποφασιστικό. Η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία τη έκφραση όσον αφορά τον πιανίστα, αυτόν τον μουσικό, τον Φαζιρσάη για παράδειγμα, είναι σημαντικά στοιχεία και πρέπει να μπορέσουμε να πούμε και να δούμε ότι είναι σημαντικό το πρωτόκολλο τη Άγγελα και συναφή θέματα να μπορέσουν να προχωρήσουν και να ευδοκιμήσουν. Και από πλευρά ε, τη Επιτροπή θέλω να προχωρήσουν αυτά. Πρέπει να γνωρίζει επίσης η Τουρκία ότι θέτουμε όρους και προϋποθέσεις χωρίς να υπαναχωρούμε για να γίνει κάποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία. Πρέπει να σέβεται αυτές τις αρχές και νομίζουμε ότι έτσι μπορεί να προχωρήσει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Ελμαμπρόκ. Για δυόμιση λεπτά ο κύριο Ρούτσεκ θα λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, Επίτροπε, συνάδελφοι. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση έρχεται σε μια σημαντική στιγμή. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη υπάρχει μια δυνατότητα για πραγματική πρόοδο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Σειρά σημαντικών και θετικών στοιχείων τελικά πηγαίνουν, μπαίνουν στη θέση τους. Πρώτα απ' όλα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις επιτέλους έχουν ε, ξεπαγώσει μετά από δύο χρόνια ένα κεφάλαιο η περιφερειακή πολιτική έχει ανοίξει και περισσότερα κεφάλαια θα πρέπει να ανοίξουν το ταχύτερο δυνατόν. Δεύτερον, νομίζω ότι το θετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη υπάρχει σαφής πρόοδος προς την Συμφωνία Επανεισδοχής καθοδόν προς την απελευθέρωση αποθεωρήσεις. Τρίτον, δίκαιη μακροχρόνια διευθέτηση του κουρδικού ζητήματος θεωρώ ότι είναι κάτι εφικτό και αν συμβεί αυτό δεν θα έθετε μόνο τέρμα σε τραγικό και βίο κεφάλαιο της τουρκικής ιστορίας αλλά θα επηρέαζε θετικά και την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας και βεβαίως θα αυξανόταν και η περιφερειακή ασφάλεια και αναφέρομαι στη Συρία πολλά απομένουν να γίνουν ε, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια ευκαιρία να συνταχθεί ένα νέο δημοκρατικό σύνταγμα. Αυτή είναι κρισίμου σημασία διαδικασία. Το δημοκρατικό μέλλον για το, το, για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας και για τη θέση της στην Ευρώπη. Άρα αυτή η συνταγματική διαδικασία μπορεί να βελτιώσει και την εδραίωση της δημοκρατίας, τη συμπερίληψη όλων, αλλά κυρίω να γίνει κοσμικό κράτος η Τουρκία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει που έχει αναλάβει και η Ευρώπη. Καμιά φορά μιλάμε για κεφάλαια 23, 24, κράτο δικαίου, δικαστικό τομέα, θεμελιώδη δικαιώματα. Μακάρι να ανοίξουν αυτά τα κεφάλαια. Μιλάμε για ενέργεια και άλλο κρίσιμο σημείο και για την Τουρκία, αλλά πάνω απ' όλα κρίσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξει και αυτό το κεφάλαιο και ε, υπάρχουν τομείς όπου θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία. Όταν μιλάμε για στατηγικά θέματα, θέματα ασφαλείας, κοιτάξτε τι συμβαίνει στη Συρία, τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία είναι κρίσιμος εταίρος, είναι προς όφελος αμοιβαίο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκία η συνεργασία. Και ξανά θα ήθελα στενότερη συνεργασία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και συγγνώμη πακριβώσα. Σα ευχαριστούμε Λίμπορ. Για 1,5 λεπτό έχετε τώρα δυνατότητα να παρέμβετε. Εσείς συνάδελφε και φίλε Άντριο Ντάφ παρακαλώ. Uh, the... Νομίζω ότι το κουρδικό πρόβλημα αν πραγματικά θέλουμε να επιληθεί πρέπει να συνδεθεί πραγματικά με μια συνταγματική μεταρρύθμιση στην Τουρκία. Αλλαγή του υπερκεντροποιημένου κράτους όσον αφορά την εξουσία στην σημερινή τουρκική δημοκρατία, τις δομές εξουσίας. Αυτό σημαίνει μεταφορά εξουσιών από την Άγκυρα σε τοπικές και περιφερειακές αρχές και κοινότητες στις τοπικές κυβερνήσεις, ακόμα και την εκλογή περιφερειακών κυβερνήσεων, επαρχιακών κυβερνήσεων. Θα πρέπει να εξεταστεί αυτή η ε, διαδικασία της αποκέντρωσης και να εμβαθύνουμε σε αυτήν. Θα πρέπει να ζητήσουμε και να ερωτήσουμε αν πραγματικά είναι συμβατή αυτή ως πρωτοβουλία με τον προφανή πρόδειλο, με την πρόδειλη επιθυμία του κυρίου Ερντοάν να μετατρέψει την Τουρκία, να την μεταμορφώσει σε ένα προεδρικού χαρακτήρα ε, καθεστώς ως ε, δημοκρατία. Υπάρχει μια συμπεφωνημένη συνταγματική διαδικασία συμφιλίωσης που ε, βρίσκεται υπό εξέλιξη και θα ήταν πραγματικά κρίμα αν σε σχέση με την, τις θέσεις του Πρωθυπουργού με μηνύματα αυταρχικά τα οποία όλο και περισσότερο εκφράζονται αυταρχικών τάσεων θα ήταν κρίμα αν αυτά όλα διακύβευαν αυτό το εγχείρημα αυτό το ιδιαίτερα ευάλωτο, περίπλοκο και σύνθετο συνταγματικά εγχείρημα των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων υπό εξέλιξη. Ευχαριστώ. Muchas gracias, Andrew. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ, Άντριο. Για ένα λεπτό τώρα, ο συνάδελφος Ντεμεσμέκερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι όλα αυτά τα προβλήματα σε σχέση με την ΕΕ και την Τουρκία πρέπει να πούμε ότι οι λύσεις αυτών των προβλημάτων βρίσκονται ως κλειδιά στα χέρια των Τούρκων. Υπάρχει και ο κίνδυνος η Άγκυρα μονομερός να θέσει όρους και προϋποθέσεις για την ειρηνευτική διαδικασία με τους ε, Κούρδους. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα σε σχέση με τις ειδήσει και τα μαντάτα για τον Οτσαλάν και τα όσα προαναγγέλλονται. Και πρέπει εδώ σε σχέση με αυτά τα οποία πρέπει να επεξηγηθούν προ του ε, πολίτε μας κάνουν πολλές φορές να διαρωτηθούμε τι συμβαίνει ακριβώς. Εκλέγονται, δηλαδή, ωραία, εντάξει, όταν εκλέγεται κάποιος στην Τουρκία ε, μπορεί να ε, ασκήσει ε, κάποια αξιώματα. Όμως ε, δεν είναι δυνατόν ως δημοσιογράφος να ασκήσει τα δικαιώματά του. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης χρήση σε σχέση με αυτά τα προβλήματα των διαπραγματεύσεων ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Κούρδοι θα έχουν πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα της γλώσσας τους, πολιτιστικά και πολιτισμικά δικαιώματα, δικαιώματα αυτονομίας, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία θρησκείας, δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης. Ευχαριστώ στην Τουρκία. Πρόεδρος, ευχαριστώ συνάδελφοι, υπενθυμίζω σε όλους να μην ομιλούν με ταχύτατο αριθμό, να ομιλούν με ένα αριθμό που θα επιτρέπουν στους διερμηνείς να παρακολουθήσουν τα όσα λέγουν και να μπορέσουν να τα διερμηνεύσουν από πλευρά τους σωστά. Για ένα λεπτό στη συνέχεια για την παρέμβασή σας, ο κύριος Ζαν Γιαχράντιλ, Ζαχράντιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω αναμφίβολα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που είναι διαφορετική από ό,τι πριν από δέκα χρόνια μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια η Τουρκία έχει γίνει μια περιφερειακή δύναμη υπό κάθε έννοια. Σήμερα το πρωί κάναμε μια συζήτηση για την Κύπρο και ο κύριος Κονμπεντίτ από την ομάδα των Πρασίνων έλαβε το λόγο σήμερα το πρωί και δεν θα φανταζόμουν ότι θα συμφωνούσα μαζί του, αλλά σήμερα συμφωνούσα γιατί τα είπε πολύ σωστά. Είπε ότι εδώ έχουμε μια ευκαιρία που παρουσιάζεται για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ξεπεράσουμε ε, ε, τη διχοτόμηση του νησιού και νομίζω ότι έχει δίκιο. Υπάρχει ευκαιρία αρκεί να δούμε ότι οι πραγματικές προσπάθειες που βασίζονται στη γενεοδορία και την καλή θέληση θα πρέπει να γίνουν ε, για να καταλήξουμε κάπου μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αυτό θα φέρει θετικό οικονομικό αντίκτυπο, θα αυξήσει τις επενδύσεις και τον τουρισμό και όπως ήδη πολλοί από είπατε και ε, στα θέματα ε, φυσικού αερίου και πετρελαίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτή τη νέα θέση της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης για να προσπαθήσουμε ε, να την κάνουμε να μας βοηθήσει περισσότερο να επιλύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Η κρίση να γίνει λοιπόν ευκαιρία εδώ ας ελπίσουμε ε, ότι θα βγάλουμε κάτι χρήσιμο από αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Για ένα λεπτό στην παρέμβασή σα, ο κύριο Αλαβράκος παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω την κυρία Ρόιτεν για την έκθεσή τη, που είναι προσεκτική και τεκμηριωμένη. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να ψηφιστεί χωρί τροπολογίε και πιστεύω ότι αποτελεί επιτυχή συνέχεια των προηγουμένων εκθέσεών τη για το θέμα καθώ μέρο δεν αναφέρει ρητά μεταβολές προς το καλύτερο. παρά τη σχετική πρόοδο που εμφανίζει η τουρκία στην εκπλήρωση των οικονομικών κριτηρίων προκύπτει ότι παραμένουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων. ως προς τις σχέσεις καλής γειτονίας η τουρκική πολιτική εξακολουθεί να υπολείπεται με τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και παράλληλα παραβιάζει τις αρχές του πρωτοκόλλου της άγκυρας που δημιουργούν υποχρεώσεις στην τουρκία σχετικά με την κύπρο πρέπει να συνεχιστούν οι δράσεις της τουρκικής κυβέρνησης για τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη το δικαιακό σύστημα και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών. ιδιαίτερα τονίζεται η αδράνεια της τουρκίας σχετικά με τις υποχρεώσεις της για το μεταναστευτικό πρόβλημα και τις υποχρεώσεις ιδιαίτερα επανεισδοχής. παράλληλα η έκθεση φωτίζει θετικά στοιχεία όπως τα σχετικά με το, τουρκικό, με το κουρδικό θέμα και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και το ρόλο της ε, τουρκίας στο συριακό πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε συνάδελφε. Για ένα λεπτό για την παρέμβασή του ο κύριο Βίλι Μέγερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, ο συνάδελφο τη ομάδα, ο Τάκη, ε, προηγούμενα τοποθετήθηκε όσον αφορά την θέση τη ομάδα. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάτι που θεωρώ ότι είναι θεμελιώδου σημασία και πρέπει να αποσταλεί ένα αναμφίσιμο μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Τουρκία. Η Τουρκία ποτέ δεν θα μπορέσει να αποτελέσει μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον εξακολουθεί να έχει υπό την κατοχή τη το βόρειο τμήμα τη Κύπρου. Το τμήμα εκείνο το οποίο βρίσκεται υπό κατοχή 40.000 Τούρκων στρατιωτών. Και σε σχέση με την πολιτική ε, που ακολουθεί υποκατοχή έχοντας ε, το βόρειο τμήμα της ε, νήσου με μια πολιτική που πραγματικά υπονομεύει την πολιτισμική ενότητα της, και της τουρκοκυπριακής μειονότητας. Για μένα αυτό είναι το αναμφίσιμο μήνυμα που πρέπει να αποσταλεί με κάθε σαφήνεια και κατηγορηματικότητα. Μπορεί να είναι σταθερότητα ε, στοιχείο και συντελεστή για την περιοχή αυτή η Τουρκία. Όμω αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Έχει υποκατοχή, παράνομη κατοχή, παράνομη κατοχή τμήμα τη Δημοκρατία τη Κύπρου. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε. Κάθετα και με, πολύ, με μεγάλη σαφήνεια. ώστε να είναι σαφέ ε, τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί από την Τουρκία υπόψη σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βίλι Μάιερ. Για ένα λεπτό ο κύριο Όμπερ Μάιερ τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί ο πράσινο Ευρωβουλευτή με ένα ιδιότυπο ε, από πλευράς πρότασης ε, ε, σχήμα το οποίο υπέβαλε είπε η Τουρκία γοργά να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα υπάρξουν αυτόματα τουρκικές επενδύσεις λέει στην Κύπρο. Γεγονός είναι ότι ο αρχικός τουρκικός πληθυσμός τη Κύπρου υφίσταται τα πάνδυνα από την δραματική μετανάστευση επίκον από την Ανατολία, από την Καπαδοκία και ανατολικέ περιοχέ τη Τουρκία στην Βόρεια Κύπρο. Και σε σχέση με τι παράλληλε αυτέ ε, πολιτισμικές σχέσει μπορεί κανεί να δει τι γίνεται στην ε, ίδια τη Γερμανία, στην ίδια την Αυστρία με αυτά τα στοιχεία. Για την πολιτισμική πολιτική όταν έχουμε κατεστραμμένε εκκλησίε ε, στο κατεχόμενο τμήμα τη Κύπρου είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Κυρίε και κύριοι, είναι εφάνταστα όνειρα αυτά τα οποία διατυπώνονται. Και σε σχέση με την Τουρκία θα πρέπει να σταματήσουν να παγώσουν οι διαπραγματεύσει με την Τουρκία. Και έχουμε επί δισεκατομμύρια τα κονδύλια τα οποία δαπανώνται και εδώ θα έπρεπε να επενδυθούν αυτά στην ίδια την Κύπρο και όχι με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, για 1,5 λεπτό η κυρία Μαρία Γιαννάκου έχει τον λόγο παρακαλώ. Αδέλφου κυρία Σόουμεν, είναι πράγματι ισορροπημένη, είναι άλλωστε επί χρόνια εισηγήτρια και παρατηρεί και χαρακτηρίζει τις μεταβολές που γίνονται στην Τουρκία. Ε, Όντω υπάρχει πρόοδος και κινητικότητα, αλλά δεν είναι η Τουρκία ακόμη μια ευρωπαϊκή χώρα το πρόβλημα είναι ότι σε πολιτικό επίπεδο ενώ υπάρχει σε άλλους τομείς πρόοδος η τουρκία εξακολουθεί να αρνείται την αποδοχή του πρωτοκόλλου της άγκυρας να διατηρεί στρατεύματα κατοχής ε, στην κύπρο ε, να μην έχει αναγνωρίσει την unclos να μην αποδέχεται το δικαστήριο της χάγης. είναι λοιπόν ένα ερώτημα η πρόοδος που έχει γίνει σε σχέση με το παλιό καθεστώς των κεμαλικών αν μπορούμε να το πούμε έτσι αντικατοπτρίζεται στις εξωτερικές της σχέσεις; η πραγματικότητα είναι όχι. δεν υπάρχει καμία κινητικότητα ουσιαστική στις εξωτερικές της σχέσεις και το λέω εγώ που εκπροσωπώ μια χώρα που θέλει την τουρκία ως μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης. τι μπορεί να κάνει η ευρωπαϊκή ένωση; δεν μπορεί να συναλλάσσεται με μια χώρα που λέει πως δεν την αναγνωρίζει ολόκληρη. είδαμε τι έγινε στην κυπριακή προεδρία. δεν μπορεί να παριστάνουμε τους αδαείς και τους αφελείς περιμένοντας ότι θα διορθωθούν αυτά με τον χρόνο. αυτά διορθώνονται μόνο υπό πραγματική πίεση. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ συνάδελφε. Για ένα λεπτό τώρα στη συνέχεια κύριος Ρίτσαρτ Χάουιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καλωσορίζει τον πακέτο που κάνει την Τουρκία να πλησιάζει περισσότερο τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά υπάρχει και η υπόθεση του κυρίου Φασίλ Σέι, κλασικού πιανίστα και συνθέτη, ε, που ε, καταδικάστηκε σε 10 μήνε με αναστολή για ένα σχόλιο το οποίο έκανε στο Twitter. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, αυτό αποτελεί μία ε, σοβαρή προειδοποίηση ότι οποιοδήποτε θέλει να εκφράσει απόψει που δεν αρέσει αρέσουν στις αρχές στην Τουρκία μπορεί να τιμωρηθεί. Επίση, υποστηρίζω διάφορε τροπολογίε που αφορούν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα αλλά και πάλι υπάρχουν απειλέ ε, κατά των ε, ε, ατόμων που ασχολούνται με συνδικαλιστικά θέματα. Μόλι πριν από δύο εβδομάδε έγιναν και όχι μόνο τώρα αλλά και στο παρελθόν υπήρξαν τέτοιε αντιπαραθέσει γύρω από την πλατεία Ταξίμ. Πρέπει λοιπόν η τουρκική κυβέρνηση να αποφύγει τέτοιε διενέξει. Υποστηρίζω τέλο την τροπολογία των σοσιαλιστών να κληθούν δύο πολίτε από την Βόρεια Κύπρο που θα αποτελέσουν παρατηρητέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητώ από ε, τους συναδέλφους να υποστηρίξουν αύριο την τροπολογία του. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε Ρίτσαρτ. Για ένα λεπτό τώρα στη συνέχεια ο κύριος Καζάκ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαίρω την κυρία Ομερόιτεν για την ισόρροπη αυτή προσέγγιση σε σχέση με την έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας Έχω την βεβαιότητα ότι η προοπτική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διέπει αυτό το εγχείρημα. Γι' αυτό οι φιλελεύθεροι καλωσορίζουμε το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 καθώς επίσης και το κεφάλαιο 15. Εμένουμε και επιμένουμε να συμπεριληφθεί η Τουρκία στις διαπραγματεύσεις ελευθέρου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών. Είναι επιτέλους η χρονική στιγμή τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσουμε σε σχέση με τους Τουρκοκυπρίους και να δοθούν και τέλος, σε σχέση με τη δυνατότητα να συμμετέχει αυτή η συνιστόσα και στις συναντήσεις ε, του Συμβουλίου. Απευθύνω έκκληση να υποστηριχθούν αυτά τα αιτήματα, ώστε να δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρεί την αρχή της ε, ενότητας ε, μέσα από διαφορετικότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, για ένα λεπτό, στη συνέχεια ο κύριος Αραμπίλαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση που υποβάλλει είναι κέρια σημασία και λέει ότι η Τουρκία έχει επιτύχει πρόοδο που θα επιτρέψει το άνοιγμα και άλλων σημαντικών κεφαλαίων στι διαπραγματεύσει και νομίζω ότι είναι σημαντικό βήμα στη διαδικασία ε, ένταξη. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα τη προστασία ε, των δικαιωμάτων ελεύθερη έκφραση και των μέσων ενημέρωση και να επιτρέπεται ελεύθερη δραστηριότητα σε διάφορε θρησκευτικέ ομάδε. Ε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την σταθεροποίηση τη κατάσταση με την έναρξη πολιτικών συζητήσεων με την κουρδική μειονότητα και θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλου τομεί και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν εγγυήσει για τα δικαιώματα και τι ελευθερίε. Και θα πρέπει να εξετάσουμε το ρόλο τη Τουρκία ω σταθεροποιητικού παράγοντα στην ευρύτερη περιφέρεια. Η δέσμευση τη Άγκυρα υπέρ τη ειρήνη και τη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή είναι ζωτική σημασία και για μα και θα πρέπει να σημειώσουμε τον ρόλο κλειδί που μπορεί να παίξει η Τουρκία στην παροχή εναλλακτικών ενεργειακών λύσεων για την Ευρώπη πέραν των, της λύσης της Ρωσίας. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε Αδάμ. Για ένα λεπτό στη συνέχεια ο κύριος ε, Κόμις του Ντάρτμουθ. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση φαίνεται τουλάχιστον εν μέρη να θέτει ε, σε αμφιβολία τα κριτήρια για την ένταξη της ε, Τουρκίας, όπως και άλλοι συνάδελφοι το έχουν πράξει. Συμφωνώ. Και ε, επειδή υπάρχουν σημαντικά ερωτηματικά για το θέμα της ένταξης της Τουρκίας, η λογική είναι ότι η προενταξιακή χρηματοδότηση προς την Τουρκία, που είναι 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2007 μέχρι το 2013, θα πρέπει να διακοπεί και να διακοπεί άμεσα. Η Τουρκία είναι ήδη στην Τελωνιακή Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ήδη αποκομίζουν όλα τα ωφέλη από το εμπόριο με την Τουρκία, όλα τα ε, ε, ωφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν. Η Τουρκία είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι ορισμένα κράτη-μέλη είναι σε στρατιωτική συμμαχία με την Τουρκία. Το γεγονός είναι ότι δεν χρειαζόμαστε την Τουρκία σε μια πολιτική ένωση. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κύριε Ντάρτμουθ. Ευχαριστώ Ρίτσαρτ. Δεν υπάρχουν εδώ μπλε κάρτες για αυτούς που παρεμβαίνουν σε αυτή τη συζήτηση. Για ένα λεπτό κύριε κύριος Σα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην πρόταση ψηφίσματος αναφέρεται ως παράθυμα η πρόοδος της Άγκυρας σε σχέση με τα δικαιώματα τα συνδικαλιστικά απαιτείται να διασφαλιστεί τέλος του παραθέματος. Και πραγματικά αυτό είναι ο εφημισμό του έτους θα έπρεπε να υπάρχει σαφήνεια σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μεγαλύτερη σαφήνεια. Δηλαδή να λέγεται ότι τα δικαιώματα των συνδικάτων καταπιέζονται και παραβιάζονται στην Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια είχαμε μια ολόκληρη σειρά διαδηλώσεων και απεργιών. Και η αστυνομία τι έκανε. Η αστυνομία βία στράφηκε κατά των διαδηλωτών και υπήρξαν και προσφυγές στα, ε, ε, προσήχθησαν στα δικαστήρια. Όλα αυτά είναι παράδεικτα. και εγώ και μια σειρά συναδέλφων έχουμε τροπολογίες που έχουμε καταθέσει σε σχέση με αυτό το ψήφισμα. Πρέπει τους όρους και προϋποθέσεις να διατυπώσουμε ώστε η Τουρκία πλήρως και απόλυτα να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Διεθνούς Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα να τα σέβεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια για ένα λεπτό ο κύριος Φιλίπ Κλές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα από πλευράς μου να πω είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο όταν ελήφθη απόφαση το 2004 να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τουρκίας μια, μιας μη ευρωπαϊκής χώρας, εννιά χρόνια αργότερα εξίσου απίστευτο είναι ότι συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Την χάνει συνέχεια. Παρόλη την απειλή ότι θα πάγωναν αυτά αν δεν υλοποιούσε η Τουρκία τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί, τους όρους και τις προϋποθέσεις. Δεν έχει νόημα να συζητάμε για έκθεση πρόοδου όταν δεν υπάρχει καμία πρόοδο να αναφέρουμε ότι σημειώθηκε στην, στην Τουρκία. Υπάρχουν περισσότεροι δημοσιογράφοι φυλακισμένοι στην Τουρκία από ότι οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Σε όλε τι άλλε χώρε. Και φυλακίζονται επειδή εξέφρασαν μια άποψη, μια γνώμη. Και ένας πασίγνωστος πιανίστας ε, του επευλήθη πίνη επειδή άσκησε λέει επίκριση στο Ισλάμ και η κυβέρνηση Ερντογάν τι κάνει. Όλο και περισσότερο γίνεται αυταρχική κατά των χριστιανών, κατά τη Δύση, κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τερματίσουμε επιτέλου αυτέ τι διαπραγματεύσει για την ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έστω για μία φορά, να λάβετε υπόψη τα συμφέροντα και τι απόψει των ψηφοφόρων τη Ευρώπη που έχουν περισσότερο μυαλό και κοινή λόγια. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια Σνίβερ Γιάστραμ. Η κυρία Σνίβερ Γιάστραμ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στην κυρία Ρία Όμεν Ρόιτεν για αυτή την έκθεση που μας δείχνει για άλλη μια φορά πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Τουρκίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο οικονομικά, ως ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, αλλά και πολιτικά. Ένας κρίκος που συνδέει την ΕΕ με την Κεντρική Ασία την ε, Ασία, τη Μέση Ανατολή. Έχει σημειώσει πρόοδου τα τελευταία χρόνια η Τουρκία σε πολλού τομεί και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Ένα από αυτού του τομεί είναι ο τομέα των μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό σκέλο. Προστοχεύει προ την σωστή κατεύθυνση. Παρόλα όσα ανέφερε ο κόμι Λάμστοφ, υπάρχουν πολλά που πρέπει να καλύψουμε. Μεγάλη πορεία που πρέπει να καλυφθεί. Και θα πρέπει ω αρρωγό να συνδράμει την Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση προ ίδιο συμφέρον τη. Γι' αυτό υποστηρίζουμε όχι μόνο τα θέματα δικαιοσύνη που πρέπει να μπορέσουν να ανοίξουν και να εξεταστούν, αλλά από κοινού θα πρέπει να αναζητήσουμε περαιτέρω τομεί όπου νέε πρόοδοι θα μπορέσουν να επιτευχθούν. Για παράδειγμα θέλω να αναφέρω τι διαπραγματεύσεις σε σχέση με το ενεργειακό κεφάλαιο. Η Τουρκία για την ΕΕ υπόσχεται πάρα πολλά ω εναλλακτική λύση έναντι τη Ρωσία. Εδώ φαίνεται ότι δεν έχουν κατανοήσει πολύ πόσο σημαντική είναι μια συνεργασία μεταξύ τη ΕΕ και τη Τουρκία στον ενεργειακό τομέα για το μέλλον. Ποια σπουδαιότητα έχει αυτό ο ενεργειακό τομέα για το μέλλον, για την ΕΕ. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στι κοινέ μα σχέσει με την Τουρκία είναι τα θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων βρίσκονται αντιφάσκοι στο πνεύμα της Τελωνιακής Ένωσης. Επιχειρηματίες αλλά και επιστήμονες αλλά και φοιτητέ να πρέπει διαρκώς κάθε φορά να ετούνται θεώρηση διαβατηρίου κάθε φορά που θέλουν να μεταβούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ολοκληρώνοντας με μια παράκληση θέλω να κλείσω. Η Τουρκία θα πρέπει δίκαια να αντιμετωπιστεί όπως και οι άλλες υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Χωρίς προκαταλήψεις, χωρί προσβολές, με τη σύνεση και την αντικειμενικότητα που πρέπει ένα Ευρωκοινοβούλιο να εκφράζει σε σχέση σχέση με ένα τέτοιο ζήτημα όπως εδώ με την Τουρκία. Η κυρία Μαριλένα Κοπά παρακαλώ έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μια ακόμα φορά συζητάμε την έκθεση προόδου για την Τουρκία. Και για μια ακόμα φορά τονίζουμε το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην ασφάλεια και ευημερία της Ένωσης. Τονίζουμε το τεράστιο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να έχει στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης αυτή η χώρα φιλοδοξεί να παίξει κεντρικό διαμεσολαβητικό ρόλο στις συγκρούσεις στη νότια γειτονιά της. μια χώρα λοιπόν που θέλει να είναι μεγάλη περιφερειακή δύναμη χθε παραβίασε για μια ακόμα φορά με τέσσερα μαχητικά αεροπλάνα τύπου f 4 και f 16 τον ελληνικό εναέριο χώρο μεταξύ των νήσων σάμου και χιου όπου και παρέμειναν για πάνω από 15 λεπτά. αυτή είναι μια καθημερινή πρακτική της τουρκίας και η καθημερινότητα των κατοίκων των ελληνικών νησιών. η ίδια η χώρα δεν δείχνει να μπορεί ακόμα να παρέχει στους πολίτες της την προστασία της ελεύθερης έκφρασης αλλά και την προστασία θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με το φετινό ψήφισμά του ζητάει για άλλη μια φορά από την τουρκία τα αυτονόητα δηλαδή σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα προστασία των μειονοτήτων βελτίωση των διμερών σχέσεων με τους γείτονές της η τουρκία δεν έχει πια δικαιολογίε. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια για ένα λεπτό ο κύριος Φαντάλεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τον προηγούμενο μήνα μόλι, ένα Τούρκο υπουργό ε, ζήτησε να υπάρξει ε, μια ε, επιστροφή όσον αφορά την Τουρκία σε αυτά. Φαίνεται ότι εδώ έχουμε μια νομική αντιπαράθεση σε σχέση με την κυβέρνηση Ερντογάν, την αντιπαράθεση σε σχέση με μοναστήρια που έχει αναλάβει η κυβέρνηση Ερντογάν. Η κατάσταση σε σχέση με τους χριστιανούς είναι απογοητευτική. Πολλοί έχουν εγκαταλείψει την Τουρκία. Εκκλησίες μετατρέπονται σε τεμένη, σε τζαμιά. Σε πρόσφατα έγινε αυτό στη Σμύρνη, για παράδειγμα. Και θα συμβεί και στην Κωνσταντινούπολη. Και έχει προαναγγελθεί ήδη αυτό από ένα δικαστήριο, δικαστή της, ε, της, της Κωνσταντινούπολης. Αν μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ερντογάν και ΠΚΚ σε σχέση με τους Κούρδους δηλαδή αυτή, αν δεν υπάρξει συμφωνία θα είναι σοβαρότατο το πρόβλημα στην νοτιοανατολική Τουρκία θα βρεθούν μεταξύ σφύρας και άκμονος οι κάτοικοι αυτών των ε, περιοχών το Συμβούλιο τώρα και η Επιτροπή έχουν πραγματικά ευθύνε όταν γίνεται λόγος για αυτά τα θέματα Πρόεδρο σας ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος ε, Ματέος Σαλβίνη Ευχαριστώ Πρόεδρε είναι σαφές ότι η Τουρκία δεν είναι και ποτέ θα μπορέσει να είναι Ευρώπη. Για λόγους ιστορικούς, για λόγους γεωγραφικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και για το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμό των δικαιωμάτων γυναικών και των θρησκευτικών μειονοτήτων, εθνοτικών, γλωσσικών μειονοτήτων. Αυτό το κοινοβούλιο μιλά για ανθρώπινα δικαιώματα κάθε τέταρτο. Και τώρα και μου έρχεται να πω ότι το αέριο και η ενέργεια μετράνε περισσότερο από την έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ θα ντρεπόμουν αν ήμουν αυτά τα άτομα που λένε αυτά τα πράγματα. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι μια υπεραγορά σούπερ μάρκετ η Ευρώπη. Ένα discount που γίνονται εκτόσει, όπου πολλούν, αγοράζουν, γίνεται ανταλλαγή προϊόντων. Αν είναι αυτό, α ανοίξουμε την Ευρώπη στον τον κόσμο. Αν θεωρεί ότι η Ευρώπη, αυτό είναι το θέμα τη Λέγα και των κατοίκων τη παδάνεια και όχι του PDL δυστυχώ σε επίπεδο ιταλικό. Αν κανεί πιστεύει ότι η Ευρώπη είναι κάτι ομοιογενέ, ε, συμπαγή, ανοιχτή, που σέβεται πράγματα, είναι υπερήφανη, η Τουρκία δεν μπορεί να είναι ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο Ευρώπη. Το μόνο λογικό για να αποφύγουμε άλλα 20 χρόνια αυτού της κοροϊδίας είναι να ανασταλούν για πάντα αυτές τις διαπραγματεύσεις με μια χώρα που δεν είναι κομμάτι της Ευρώπης και είναι σαφές σε όλους πιστεύω. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό θα έχει τον λόγο ο κύριος Κλούτε, παρακαλώ. Ο κύριος Κλούτε, ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, από τα τέλη του 2012 παρακολουθούμε μια ιστορική σημασία ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ της κυβέρνησης της Άγκυρας και των ανταρτών του ΠΚΚ που εκπροσωπούνται στο κυριότερο μέρος από τον ε, κύριο Τζαλάν. Έχουμε ε, μια σύραξη που εδώ και 30 χρόνια ε, ήταν ματηρή στην η σύραξη αυτή και προκάλεσε πάρα πολλά θύματα. Επί μεγάλο χρονικό διάστημα προσπάθησαν με τη βία να επιλύσουν οι Τούρκοι το πρόβλημα της βίας. Είναι καλό τώρα ότι υπάρχει αλλαγή νοοτροπίας και στις δύο πλευρές. Και τώρα σε σχέση με τον Αμπτουλά Οτσαλάν δήλωσε ότι ήρθε η χρονική στιγμή να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας, η ένοπλη σύραξη και ότι θα έπρεπε να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία. Δεν πρέπει να αφήσει καμιά αμφιβολία η Ευρώπη ότι υποστηρίζει χωρίς καμία αμφισημία ενωμένη αυτή την ε, πρόθεση, αυτή την ε, ειρηνευτική διαδικασία. Θα πρέπει εκ των έξω να δράσουμε ως διαμεσολαβητές ε, σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Όμως κάνουμε λόγο στην έκθεση για την Τουρκία, για το ΠΚΚ ως τρομοκρατική οργάνωση. Διαρωτώ με, αυτό είναι επικοδομητικό σε αυτή τη φάση που διεξάγονται ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Δεν θα έπρεπε ως Κοινοβούλιο να απόσχουμε από τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Για 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Βαλένσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, το Τουρκικό Κοινοβούλιο ενέκρινε κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αυτό είναι πολύ θετικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αυτό είναι απλώς ένα βήμα στο δρόμο που έχει να κάνει η Τουρκία για να υιοθετήσει ε, τα ισχύοντα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν δημιουργήσει ανησυχίε τα τελευταία χρόνια σχετικά με την Τουρκία ακόμη και το καλύτερο νομοσχέδιο δεν εγγυάται την τήρηση του τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά θα πρέπει ε, να ερμηνευθούν και η ερμηνεία της νομοθεσίας είναι σημαντική. Όπως βλέπουμε στην περίπτωση του κλασικού πιανίστα, ο οποίος καταδικάστηκε διότι θεωρήθηκε ότι προσέβαλε το Ισλάμ μετά από ένα μήνυμα που είχε γράψει στο Twitter και υπάρχουν ε, και παραδείγματα δημοσιογράφων που έχουν ε, φυλακιστεί σύμφωνα με τον ε, αντιτρομοκρατικό νόμο και είναι κάτι το οποίο πρέπει να θέσουμε στις τουρκικές αρχές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία και να εξετάζει τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα στην Τουρκία και να βρει εγγύησεις ότι υπάρχει η ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης Υπάρχει το κεφάλαιο για το δικαστικό σώμα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα αποτελέσει κλειδί για την πραγματική επιτυχία το να τηρούνται αυτές οι διατάξει. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, κύριο Σοφοκλέου, παρακαλώ. Επανέρχεται η συζήτηση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Είναι η ώρα να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας, σε αυτά που συμφωνούμε και μας δεσμεύουν, αλλά και σε αυτά που οφείλουμε να πράξουμε, να απαιτήσουμε, να αντιδράσουμε επίση μα δεσμεύω. συμφωνούμε ότι η τουρκία είναι σημαντικό εταίρο τη ευρωπαϊκή ένωση αλλά και πρέπει να απαιτούμε η τουρκία να σέβεται εμπράκτο την ευρωπαϊκή ένωση. αυτή είναι η προπόθεση για να βρεθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. συζητούμε για αυτά που όφιλε να κάνει προ την εκδημοκρατικοποίησή τη αλλά πιο σημαντικό είναι αυτά που δεν έκανε και όφιλε όμω να τα κάνει. η συμμετοχή τη δεν είναι la τα ανθρώπινα δικαιώματα ελευθερία του τύπου καταπνίγονται περιορίζονται φυλακίσεις σε δημοσιογράφους κούρδους πολίτες που αγωνίζονται για δημοκρατία ελευθερία συνεχίζονται με συνοπτικές διαδικασίες. η ισότητα των δύο φύλων για την ώρα είναι αδιανόητη. και βέβαια συνεχίζεται η εισβολή η κατοχή των εδαφών της κυπριακής δημοκρατίας καταπατά κάθε αρχή δικαίου. υπενθυμίζω δηλώσεις προκλητικές απαράδεκτες από τούρκους αξιωματούχους τώρα πρέπει να τις αποσύρουν να πούν τη δική τους συγγνώμη. ο πρόεδρος γκιουλ στις 23 ε, ε, εντεκάτου του 2011 αναφερόμενος για την κυπριακή δημοκρατία μια μισή χώρα θα κληθεί μιας άθλιας ένωσης. αλήθεια είμαστε άθλιοι. ο μπαγής δηλώνει ανύπαρκτη κυπριακή προεδρία της ευρωπαϊκής ένωσης. αλήθεια αυτός είναι ο σεβασμός η αναγνώριση ενός κράτους μέλους σεβασμός στην ένωση θα το αποδεχόταν κανείς από εσά για τη χώρα του. συμπερασματικά τελειώνω. η τουρκία δεν έχει μέλλον προς την ευρωπαϊκή ένωση όσο συμπεριφέρεται ας μου επιτραπεί η έκφραση σαν τρελό Πρόεδρο, έληξε ο χρόνο σα, ε, και μάλιστα τον ξεπεράσατε κατά πολύ συνάδελφε. Για 1,5 λεπτό η κυρία, η δόκτωρ Θεοχάρου, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε κατανοώ πόσο δύσκολο είναι το έργο της κυρίας Σόουμεν να συγγράψει την έκθεση αξιολόγησης της τουρκικής ενταξιακής πορείας. κατανοώ επίσης πόσο δύσκολο είναι να γίνουν συμβιβασμοί λόγω των πολλαπλών και αλληλοσυγκρουμένων συμφερόντων και λόγω του ότι δεν πριτανεύει πάντοτε στις αποφάσεις μας το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ο διεθνής νόμος αλλά ο συγκερασμός θέσεων. για παράδειγμα αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε τον τεράστιο όγκο συναλλαγών που έχει η ευρωπαϊκή ένωση με την τουρκία η τουρκία όντω έχει κάνει πρόοδο και μεταρρυθμίσει, αλλά είναι η ίδια που παρεμποδίζει την ένταξή τη. συνάδελφοι κατανοήστε και την δική μου τη θέση καθώ προέρχομαι από μια χώρα κατεχόμενη από τον τουρκικό στρατό. η τουρκία ενώ συνεχίζει την κατοχή και τι απειλέ, τώρα προβάλλει και το ζήτημα παρουσία τουρκοκυπρίων παρατηρητών στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στην πραγματικότητα κύριε επίτροπε εκείνο που επιδιώκει είναι την εκπροσώπηση του ψευδοκράτους και την προαγωγή και μονιμοποίηση της διχοτόμησης. άλλωστε οι τουρκοκύπροι μπορούν άνετα και ελεύθερα να λάβουν μέρος στις ευρωεκλογές ως πολίτες της κυπριακής δημοκρατίας. η κυπριακή δημοκρατία προστατεύει όλους τους πολίτες της και φυσικά τους τουρκοκύπριους οι οποίοι επιπλέον απολαμβάνουν προνόμια που δεν τα έχουν άλλοι πολίτες και όλα τα προνόμια που του διασφαλίζει η ιδιότητα του πολίτη τη κυπριακή δημοκρατία. συνεπώ για να φτάσει η τουρκία στην ένταξη πρέπει να σεβαστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο πρέπει να σεβαστεί το διεθνή νόμο να αναγνωρίσει την κυπριακή δημοκρατία να μην απειλεί την κύπρο και την ελλάδα να, βοηθήσει στην επίλυση του κυπριακού προβλήματο στη βάση των αρχών και των αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Κύριε Επίτροπε, η Κυπριακή Δημοκρατία δέχθηκε πέρυσι τέτοιο καιρό την θετική ατζέντα αλλά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ειδικά εσείς ποια ήταν η ανταπόκριση της τουρκίας στην ε, ε, στάση της κυπριακής πολιτείας. Κύριοι συνάδελφοι, παρά τις επιφυλάξεις μου σε ορισμένα θέματα, θα δώσω θετική αλλά αιτιολογημένη ψήφο στην έκθεση της κυρίας Όμεν ως ένδειξη σεβασμού στο πολύ δύσκολο έργο που παράγει η συνάδελφος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε Ελένη. Πολύ. Ελένη, προσέξτε. Υπάρχει ένας συνάδελφος, ο συνάδελφος Στέντλερ, ο συνάδελφος Στέντλερ, που θέλει να υποβάλει ερώτηση προς εμάς. Ελένη, τη δέχεστε αυτή την ερώτηση, ναι. Γίνεται δεκτή η ερώτηση. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, συνάδελφε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγα λεπτά ένας, μία συνάδελφος από την ομάδα σας είπε ότι πρέπει ίσα να αντιμετωπίζεται η Τουρκία όπως κάθε υποψήφια προς ένταξη χώρα. Εσείς ως Ευρωβουλευτής από την Τουρκία έχετε εξετάσει αν υπάρχει ένα προηγούμενο, ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απορρίπτει μία τέτοια ε, προοπτική όταν ε, αρνείται ε, τα επικυριαρχικά της δικαιώματα μία χώρα ή αν ένα άλλο κράτος υπήρξε ως προηγούμενο που να έχει κάνει γενοκτονία σε σχέση με την Αρμενία για παράδειγμα τους Αρμενίους και την άρνηση μιας τέτοιας γενοκτονίας. Αυτό θα πρέπει να αποσαφινιστεί για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει ίση μεταχείριση υποψήφιων προς ένταξη χωρών και αν η Τουρκία μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της ένα τέτοιο περιθώριο. Ευχαριστώ. Σίγουρα, σίγουρα η Τουρκία απολαμβάνει μια προνομιακή μεταχείριση. Νομίζω ότι όλοι το κατανοούν αυτό το ζήτημα. Σίγουρα δεν έχει συμμορφωθεί σε πολλού ρητού όρου που τη έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει εφαρμόσει την αντιδήλωση τη 21 η Σεπτεμβρίου, δεν έχει εφαρμόσει το πρωτόκολλο τη Άγκυρα και παρόλα αυτά εξακολουθεί να ε, συνομιλεί με την ευρωπαϊκή ένωση να μην αναγνωρίζει την κυπριακή δημοκρατία να μην δέχεται την κυπριακή προεδρία να απειλεί λόγης και έργης την προσπάθεια της κυπριακής δημοκρατίας να φέρει στην επιφάνεια από το βυθό της θάλασσας τον φυσικό της πλούτο και παρόλα αυτά όλοι ε, κάνουν πως δεν συμβαίνει τίποτε. είχα κάνει την ίδια ερώτηση ακριβώς και στον κύριο επίτροπο πριν από αρκετό καιρό για αυτή ακριβώς τη συμπεριφορά της τουρκίας. νομίζω επιτέλους ότι πρέπει να σεβαστούμε τις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης και όχι τον όγκο συναλλαγό που έχει η ένωση με την τουρκία. ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Θεοχάρου. Για ένα λεπτό κυρία Μπος παρακαλώ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Όμεν Ρόιτεν και να ευχαριστήσω τον κύριο και σκιώδη εισηγητή της ομάδας μας ε, για την ε, δουλειά που έχει κάνει για το ίδιο θέμα. Η έκθεση υποστηρίζει το άνοιγμα πέντε νέων κεφαλαίων διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα ότι εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να υπάρξει πρόοδο στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Η έκθεση επίσης εντοπίζει τους τομείς στους οποίους ακόμη υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Χρειάζεται σαφώς μια νομοθεσία, ναι, για διάφορα θέματα όπως για την ελευθερία της έκθεσης. Η έκθεση αυτή όχι μόνο επικρίνει την Τουρκία αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι αν πραγματικά θέλουμε βελτιώσεις θα πρέπει να αρχίσουμε πραγματικές διαπραγματεύσεις και αν αντιμετωπίζουμε σοβαρά το θέμα της υποστήριξης της επανένωσης ε, της νήσου Κύπρου θα πρέπει να βοηθήσουμε ούτως ώστε οι Ελληνοκύπροι να συμμετάσχουν στη δημοκρατική διαδικασία. Νομίζω ότι είναι είναι λοιπόν πολύ καλή ιδέα το να υποστηρίξουμε την τροπολογία που ζητεί από τον Πρόεδρο να εξετάσει τη δυνατότητα τουρκοκυπρίων παρατηρητών εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. σε ευχαριστώ Εμίν Μποσκούρτ. Για 1,5 λεπτό τώρα θα λάβει τον λόγο ο συνάδελφος Νταζόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που έκανε μια ισορροπημένη και σαφή έκθεση σε ένα δύσκολο πλαίσιο, διότι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Τουρκίας ε, τίθεται σε ένα πλαίσιο όπου δεν είναι δυνατόν να επιτελέσουμε πρόοδο χωρίς η πρόοδος αυτή να μπαίνει στην προοπτική της ένταξης. Γνωρίζουμε ότι αυτή η προοπτική της ένταξης από μόνη της είναι προβληματική. Είναι προβληματική για πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής για την κοινή γνώμη και για την Τουρκία την ίδια είναι προβληματική. Γνωρίζουμε ότι αυτή η ένταξη δεν την χάνει συνένεση. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, λοιπόν, πρέπει να θέσουμε το ερώτημα σχετικά με ε, την πρόταση ανοίγματο πέντε νέων κεφαλαίων. Γιατί, όπω ακούσαμε μόλι τώρα, είναι ένα πολιτικό μήνυμα αυτό που δίνεται. Το άνοιγμα κεφαλαίων σαφώς αποτελεί ένα μοχλό για τη βελτίωση κέριων και ευαίσθητων τομέων ε, στα θέματα που θα διαπραγματευτούμε. Αλλά πριν μπούμε στις διαπραγματεύσεις επί της ουσίας, στέλνουμε ένα πολιτικό μήνυμα, διπλό μήνυμα. Ένα μήνυμα ανταμοιβή της Τουρκίας ε, και στη τωρινή συμπεριφορά της Τουρκίας δεν βλέπω τι μας επιτρέπει να την συγχαρούμε, ιδίως βλέποντας τη στάση της προς την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δεύτερο μήνυμα που στέλνουμε είναι ένα μείνουμε προς την κοινή γνώμη στι χώρες μας ότι μπαίνουμε σε μια μηχανιστική πορεία ένταξης και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ευαισθησία του θέματος ε, των διευρύνσεων πέραν ε, του τουρκικού ζητήματος. Θα πρέπει να προσέξουμε για να μην αποπροσανατολίσουμε την κοινή γνώμη και του Ευρωπαϊκού Λαού. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Στη συνέχεια για μισή λεπτό η κυρία Ρενάτε Ζόμερ, παρακαλώ. Ναι, και εγώ θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ και την εισηγήτρια και να την ευχαριστήσω θερμά για την έκθεσή τη που είχε θετική έκβαση. Ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο είναι δύσκολο, δυσχερέ αυτό το εγχείρημα αυτού του έργου που επιτελέστηκε. Το ψήφισμα είναι συνολικά ικανοποιητικό, αλλά με πολλά στοιχεία δεν συμφωνώ. Το άνοιγμα 5 έως 6 όπως ζητείτε ε, κεφαλαίων υποδιαπραγμάτευση όπως ζητείτε είναι κάτι απαράδεκτο, απόλυτα απαράδεκτο δεδομένη της κατάστασης στην Τουρκία και δεδομένης της τάσης και τοποθέτησης της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και χρόνια ασκούνται επικρίσεις ε, για το πάγωμα των προ... της προόδου της διαπραγματεύσης και τώρα πάλι γίνεται λόγος ε, για την παραβίαση θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων. Είναι μια πιστοδρόμηση αυτή. Ταυτόχρονα η Τουρκία δείχνει ότι η ΕΕ στο σύνολό της και ως ολοκληρωμένο θεσμικό όργανο δεν αναγνωρίζεται από την Τουρκία και για την ε, ε, Τουρκία είχαμε την άρνηση έναντι της ε, Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου να την αναγνωρίσει πως είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζει η Τουρκία την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέει ότι υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση από 26 και όχι 27 κράτη-μέλη απαράδεκτο αυτό και σε σχέση με την ε, επικύρωση της Συμφωνίας Επανεισδοχής όλο και νέα αιτήματα τίθενται ε, ε, όσον αφορά την ευρωπαϊκή πλευρά από τους Τούρκους ε, για την επικράτεια της Τουρκίας ώστε να ασκηθούν πιέσεις και να δια της βίας πετύχουν διευκολύνσεις θεωρήσεων διαβατηρίων. Ναι, η Τουρκία είναι σημαντικός οικονομικός εταίρος, εμπορικός εταίρος και στις εξωτερικές σχέσεις και όσον αφορά και την ασφάλεια, σίγουρα. Εφόσον όμως η χώρα δεν υλοποιεί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπενχάγης, εφόσον αρνείται αυτή η χώρα να μετεξελιχθεί δημοκρατικά και σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τα κεφάλαια 23-24, κράτος δικαίου, δικαστικό, δικαιώματα, δεν είναι δυνατόν να μη σημειώνεται πρόοδος. Θα πρέπει εδώ να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα, διότι πραγματικά η Τουρκία δεν ε, μεταφέρει και δεν μπορεί να αφομοιώσει όλα αυτά. Και δεν είμαι υπέρ του να υπάρξει η ε, παροχή αερίου και πετρελαίου μέσω ενός αγωγού Ναμπούκο και να πουλήσουμε την ψυχή μας για αυτό. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριο Λίσεκ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα επαναλάβω και εγώ τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστήρες προς την κυρία Όμεν Ρόιτεν για την πολύ καλή αυτή έκθεση. Είναι ένα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο θέμα αλλά νομίζω ότι τα κατάφερε πολύ καλά να ανταποκριθεί στην πρόκληση που της ετέθη. Κανείς δεν θα τα είχε καταφέρει καλύτερα από εσά. Επί τη ουσία τώρα, όταν ε, ε, ακούμε τις γνώμες των εμπειρογνωμόνων και των ειδικών ε, συχνά υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις όπως και μεταξύ των πολιτικών. Η χώρα μου, η Πολωνία, υποστηρίζει τη μελλοντική ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θα ήμουν υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων για την ένταξη ούτως ώστε να έρθουν όλοι οι φραγμοί που υπάρχουν και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο άνοιγμα περαιτέρω κεφαλαίων στι διαπραγματεύσει και πρέπει να το κάνουμε ιδίω για να δείξουμε στου συναδέλφου μα στην Τουρκία και για να δείξουμε στου πολιτικού και στο τουρκικό κοινοβούλιο και στην τουρκική κυβέρνηση πού ακριβώ βρίσκονται τα προβλήματα, τι είδου είναι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, ποιε πολιτικέ είναι εσφαλμένε διότι πιστεύω ότι οι Τούρκοι πολιτικοί θα καταλάβουν ε, ε, τα σημεία στα οποία πρέπει να διορθώσουν την κατάσταση. Η κατάσταση στην Κύπρο βεβαίω είναι απαράδεκτη και από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάσουμε το πώ μπορούν να επιληθούν ω προτεραιότητα αυτά τα θέματα. για 1,5 λεπτό τώρα κύριος παρακαλώ. Πρόεδρε, δεν κατανοώ τη συμπάθεια του συναδέλφου Ζάχραντιλ για περιφερειακές ε, υπερδυνάμεις. Έχουμε αρνητική πείρα με τέτοιες ε, ε, περιφερειακές υπερδυνάμεις. Και την ιδέα του φεντεραλισμού, ενός φεντεραλισμού που τους ίσους τους κάνει λίγο μεγαλύτερους και υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Όποιος θέλει να είναι υπέρ μιας φεντεραλιστικής δομής δεν, δεν μπορεί να είναι υπέρ της ένταξης μιας μεγάλης της περιφερειακής χώρας που δεν ανήκει σε αυτή την ε, δομή. Πρέπει σε στενή σχέση να έχουμε μια εταιρική σχέση με την Τουρκία. Ναι, και η έκθεση της κυρίας Όμερ Ρόιτεν είναι πραγματικά ισορροπημένη. Όμως το να ανοίξουμε κεφάλαια τώρα με την Τουρκία που στοχεύουν στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο σε εταιρική σχέση με την Τουρκία είναι αντιπαραγωγικό και είναι παραπλανητικό. Είναι λαθασμένη πορεία. Τώρα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα Βαλκάνια, όπου πάνε τόσο μακριά ώστε σε χώρες όπως το Κωσυφοπέδιο, την Αλβανία, τη Βοσνία, Εζεγοβίνη, θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία. Και πώς είναι δυνατόν να δεχτούμε κάτι τέτοιο τουρκική περίοδος ε, αναφέρεται ότι είναι μια παραδείσια εποχή και δεν είναι δυνατόν λέει να υπάρχει κατοχή. Επιθετικά αναμειγνύονται μέσω των ε, πρέσβεων σε εσωτερικές υποθέσεις και των δύο αυτών χωρών. Και σας λέω μια τέτοια νεοοθωμανική εξωτερική πολιτική από την Τουρκία δεν ωφελεί σε τίποτα και στον πολιτιστικό πολιτισμικό τομέα δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικός εταίρος για την Ευρώπη η Τουρκία αλλά δεν είναι ούτε υπερπεριφερειακή δύναμη ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Μιγιάν παρακαλώ. Η διαδικασία ένταξης η Τουρκία έχει κάνει μια ολόκληρη σειρά μεταρρυθμίσεων οικονομικών και πολιτικών που συνεισφέρουν σημαντικά στον εξυγχρονισμό αυτή τη χώρα. Και το ίδιο γίνεται και από άλλε χώρε ε, σε σχέση με μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση θα ψηφίσουμε αύριο τη κυρία Όμεν Ρόιτεν που τη συγχαίρω, ενθαρρύνεται η τουρκική κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή τη σημαντική διαδικασία μεταρρυθμίσεων που έχει επιπτώσεις και στο ίδιο το τουρκικό σύνταγμα. Εγώ δεν ασκώ επικρίσεις για το άνοιγμα του κεφαλαίου 22 όπως προαναγγέλθηκε σε σχέση με την περιφερειακή πολιτική έκθεση Όμεν Ρόιτεν δείχνει το άνοιγμα νέων κεφαλαίων για τη διαπραγμάτευση όπως το 2015 για παράδειγμα για τα ενεργειακά θέματα. Εγώ πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ενεργειακά θέματα είναι πολύ σημαντική. Πρέπει οι Ευρωπαίοι να πολυμορφοποιήσουμε την ε, δυνατότητα ανεφοδιασμού μας σε σχέση με ενεργειακά προϊόντα. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης η Τουρκία έχει ένα στρατηγικό ρόλο, στρατηγική σημασία και λόγω αυτής της γεωγραφικής τοποθεσίας είναι αναγκαία η συνεργασία της Τουρκίας όσον αφορά και τις ροές μεταναστών, μεταναστευτικές ροές που ε, περνούν από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Και δυστυχώς δεν έχει ε, υπάρξει κάποια προσέγγιση σε σχέση με την πολιτική της Τουρκίας για τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Και ολοκληρώνω. Για μένα ο συντονισμός και ο διάλογος για την εξωτερική πολιτική μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας είναι κάτι σκόπιμο. Και για την Τουρκία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο συμβαίνει και με την Νότια Πτέρυγα, με τις αραβικές χώρες, με την ε, Βόρεια Αφρική έχουμε εδώ ε, γείτονε που σε σχέση με μια μεγάλη περίοδο μεταρρυθμίσεων έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να συντονιστούμε ιδιαίτερα Τούρκοι και Ευρωπαίοι ώστε τα μηνύματα αυτά προ του γείτονε να περνάνε προ μια ενιαία κατεύθυνση υπέρ τη ε, ευημερία, τη ελευθερία ε, και τη ανάπτυξη του. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ κύριε Μιγιάν. Τελευταίο αγορητή σε αυτό το γύρο είναι ο κύριο Πέτερλε. Έχει 1,5 λεπτό παρακαλώ για την παρέμβαση του κύριος Πέτερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Στην έκθεση της κυρίας Όμεν Ρόιτεν καλύπτεται το θέμα της πρόοδου της Τουρκίας και αναγνωρίζω ότι είναι μια ισορροπημένη έκθεση. αναγνωρίζει την πρόοδο, καταδικάζει, ανησυχεί. Αυτά αναφέρει η έκθεση στις διάφορες παραγράφους. Μιλάμε για ενδυνάμωση του πολιτικού διαλόγου με την Τουρκία και γνωρίζουμε ποια είναι τα σημεία που πρέπει να επικρίνουμε. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων και λαμβάνοντα υπόψη όλε τι διαφωνίε που ακούσαμε και σήμερα, πιστεύω παρόλα αυτά ότι έχει νόημα το να ανοίξουμε νέε διαπραγματεύσει ε, για να μπορέσουμε να εργαστούμε για το αμοιβαίο συμφέρον, ιδίω όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την ενεργειακή πολιτική. Υπάρχουν πολλά ζητήματα όπου δεν χρειαζόμαστε νέα πλαίσια ή νέε συνθήκε, αλλά παρά μόνο καλή θέληση. Σε ευχαριστώ Αλόης. Ολοκληρώσαμε τον γύρο των αγοριτών. Περνάμε τώρα στο Catch the Eye από πλευρά Προέδρου που θα δώσει τον λόγο σε ευρωβουλευτέ. όπω πάντα έχουμε πάρα πολλού περισσότερου αγορητέ που ζητούν να παρέμβουν σε σχέση με τον χρόνο που είναι διαθέσιμο. Θα προσπαθήσω να δώσω τον λόγο σε όλου, έχοντας αποκαταστήσει κάπως το ωράριο. Αλλά να λάβετε υπόψη ότι όπως πάντα, μόλις θα ολοκληρωθεί το λεπτό, θα αφαιρώ τον λόγο από τον αγορητή. Θα αφαιρώ το μικρόφωνο. Πρώτος,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 Πρόεδρος, ε, τώρα θα λάβει τον λόγο η κυρία Παπαδοπούλου παρακαλώ. Mr. President. Mr. Κύριε Πρόεδρε, κύριε κύριος και ο κύριος Κονπεντήτ φαίνεται ότι αγνοούν ότι η Τουρκία, υποψήφια προς ένταξη χώρα, συνεχίζει ε, να έχει σε παράνομη κατοχή το 37% του εδάφου της Τουρκίας επί 39 έτη, παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο για άλλη μια φορά κάνω έκκληση ε, προς εσάς να στείλετε ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι αν επιθυμεί την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις της σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει καλές σχέσεις καλής γειτονίας, να εφαρμόζει το πρωτόκολλο της Άγκυρας, να αναγνωρίσει τη δημοκρατία της Κύπρου ως κυρίαρχο ε, ε, κράτος με μια ηθαγένεια για τους πολίτες. Είναι απαράδεκτο το να συζητούμε τροπολογίες για χορήγηση καθεστώτος παρατηρητού σε πολίτες της Βορείου Κύπρου γιατί αυτό θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τη συνθήκη είδηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι απαράδεκτο να ανοίξει νέο κεφάλαιο. Διακόπτεται. Αφαιρέθηκε το μικρόφωνο. Thank you, President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 προηγούμενη έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας σημειώνουμε ότι υπάρχουν σημαντικές πρόοδοι και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό τομέα και σε άλλους τομείς όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της οικογένειας. Αλλά οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν ένα πολύ μικρό βήμα προς τα εμπρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει την Τουρκία για να συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή διότι υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου χρειάζονται ριζικές μεταρρυθμίσεις. Η μεταρρύθμιση του συντάγματο είναι μια θετική εξέλιξη και ολόψυχα ελπίζω ότι θα υπάρξουν θετικέ πρόοδοι ούτω ώστε το σύνταγμα να είναι ε, σύμφωνο με τα κριτήρια τη Κοπεχάγης διότι θα πρέπει να υπάρχει διάκριση των εξουσιών στο κράτο και διάκριση μεταξύ κράτου ε, και ε, θρησκείας και εγγύηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαιρετίζω τι θετικέ εξελίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτω ώστε να ανοίξουν νέα κεφάλαια για τι διαπραγματεύσει. Πιστεύω ότι θα πρέπει... Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε συνάδελφε. Εξαντλήθηκε ο χρόνο σα. Ο κύριο Βλάσακ παρακαλώ. Αγαπητέ Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το μέγεθος της αγοράς και όσον αφορά και θέματα πολιτικής ασφάλειας, η Τουρκία είναι ένας εταίρο πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι η διαδικασία ένταξη αποτελεί μία από τις καλύτερες ευκαιρίες για να υποστηρίξουμε ε, τις μεταρρυθμίσει τις οποίες εφαρμόζει η Τουρκία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιώματα των γυναικών, και ούτω καθεξής. Ε, θα πρέπει ε, να έχουμε κατά νου ότι η Τουρκία είναι ο έκτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η Τουρκία ε, για τη δημιουργία των οδών διαμετακόμισης στον ενεργειακό τομέα. Θα πρέπει να εξετάσουμε θετικά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας όπως επίσης και τις μεταρρυθμίσεις του συντάγματος θα πρέπει να θέσουμε προς το Κυπριακό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπάτεν έχει τον λόγο παρακαλώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γιατί θέλει η Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχήν. Φαντάζομαι ότι θέλει να υποφεληθεί από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις όπως τόσες χώρες πριν από την Τουρκία. Ως σχετικά φτωχή χώρα φαντάζομαι ότι η Τουρκία επίσης ελπίζει ότι θα στείλει κάποιους από τους πιο φτωχούς ε, πολίτες της από το ε, κράτος με τον υπερπληθυσμό που έχει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ανοιχτών συνόρων, της πολιτικής ανοιχτών συνόρων τον όρο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία έχει 73 ε, εκατομμύρια κατοίκου και πολλοί από αυτού φαντάζομαι να ανοίξουν τα σύνορα θα φτάσουν και στη Βρετανία. Φαντάζομαι ότι θα έρθουν είτε για να δουλέψουν είτε για να υποφεληθούν από το σύστημα στέγαση ε, και πολιτικών ε, επιδομάτων ανεργία όπω πολλοί πριν από αυτού υποφελήθηκαν. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα συντηρητικά και εργατικά, το συντηρητικό και το εργατικό κόμμα είναι υπέρ τη ένταξη τη Τουρκία ανοίγοντας το δρόμο σε μεγαλύτερη μαζική ε, μετανάστευση. Ευχαριστώ κύριε Μπάτεν. Ο κύριος Τενταφυλίδης έχει το λόγο. Πρόεδρε, επειδή έχουν ακουστεί φωνές υπέρ του ανοίγματο του κεφαλαίου για την ενέργεια, καθώς και της εκπροσώπησης των τουρκοκυπρίων στο Ευρωκοινοβούλιο, θέματα που εκ πρώτη όψεω πιθανόν να ακούγονται σωστά και δίκαια, θα ήθελα να εξηγήσω γιατί αυτέ οι προτάσει, σε περίπτωση που ήθελαν να υιοθετηθεί, θα καταστρατηγούσαν βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, υπενθυμίζουμε ότι η αρχή τη κυριαρχική ισότητα των λαών είναι βασική αρχή λειτουργία τη Ένωση ω εκ τούτου δεν μπορεί το ευρωκοινοβούλιο να υποστηρίζει το άνοιγμα του κεφαλαίου τη ενέργεια όταν η υποψήφια για ένταξη χώρα επιμένει να καταστρατηγεί το σχετικό διεθνέ δίκαιο που είναι και ευρωπαϊκό. δεύτερον όσον αφορά το θέμα τη εκπροσώπηση των τουρκοκυπρίων στο κοινοβούλιο εκτιμούμε ότι πρόκειται για μια θέση που ενθαρρύνει όσου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα επιδιώκουν λύση δύο χωριστών κρατών. η κυπριακή δημοκρατία δεν έχει στερήσει στι ευρωεκλογέ από όποιο πολίτη τη Κύπρου, Ελληνοκύπριων ή Τουρκοκύπριων, το δικαίωμα του εκλέγεν και εκλέγεστε. Ε, τελείωσε ο χρόνος ομιλίας σας. Επόμενος ομιλητής, κ. Μπρόγκς. Ε, σαφώς υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν η Τουρκία καταδικάζει τους ακαδημαϊκούς για την έκφραση της, ε, της γνώμης τους όπως ε, το ότι χαρακτηρίζουν τη δολοφονία των Αρμενίων ως γενοκτονία καταδικάζονται ε, ε, ε, στη Γαλλία επίσης αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν ήταν γενοκτονία. Ίσως τελικά λοιπόν η Τουρκία να μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού το ίδιο κάνουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα προτιμούσα να είμαι περισσότερο ευρωπαϊκός παρά λιγότερο φιλοευρωπαίος όσο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα θα ήθελα να υπάρχει. Η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκό κράτος μέλος ούτε από τη γεωγραφία, ούτε από την κουλτούρα, ούτε από την ιστορία. Πιστεύω ότι μια χώρα που συνεχίζει συνεχίζει να κατέχει σχεδόν 40% της Κύπρου μπορεί ακόμη να θεωρείται ότι μπορεί να είναι υποψήφια για να γίνει μέλος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Δεν βλέπω τον κύριο Μίλτο στη θέση του. Είχε ζητήσει το λόγο, αλλά νομίζω τώρα ολοκληρώσαμε με τη διαδικασία Catch the Eye. Και επομένως μπορούμε να περάσουμε στο τελευταίο τμήμα της συζήτησης αυτής. Ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει το λόγο ο Επίτροπος Φιούλε. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υπουργέ, αξιότιμα μέλη, δεν είναι η πρώτη φορά που είχα το προνόμιο να συμμετάσχω σε αυτή τη σημαντική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα, συνεπώς, ως σκέψη, να πω τα εξής δύο πράγματα. Πράγματα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτή η συζήτηση σαφώς δείχνει ότι αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε πλήρης ενότης μεταξύ μας όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο ζήτημα. Πράγματι, δύσκολο να κρίνει κανείς το σήμερα. Πέρασαν πολλά χρόνια από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. για πολλούς και διαφόρους λόγους είμαστε ακόμα στην αρχή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Τα 13 κεφάλαια από τα 13 πάνηξαν μόνο ένα έκλεισε προσωρινά. Είμαι βέβαιος ότι θα έρθει η στιγμή και πρέπει να εργαστούμε γι' αυτό. Θα έρθει η στιγμή που θα μπορέσουμε να κάνουμε την αποτίμηση, να κρίνουμε, έχοντας από τη μία πλευρά την Τουρκία που θα περάσει από όλα αυτά τα 35 κεφάλαια, ανταποκρινόμενες υποχρεώσεις της, και από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να δώσει στα κράτη-μέλη σαφή αξιολόγηση του αντίκτυπου που θα είχε η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτεραιότητα δεν είναι να συγκεντρωθούμε επί υποθετικών ζητημάτων τώρα. Αν θα έχουμε τα πάντα στο τέλος της διαδικασίας. Ας επικεντρωθούμε τώρα στη διαδικασία αυτή κάθε αυτή. Ας ενισχύσουμε την αξιοπιστία της. Αξιοπιστία και από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευρά τουρκικής πρέπει να ενισχυθεί. Η αξιοπιστία από πλευρά τουρκική, τι εννοώ δηλαδή. Να γίνουν μεταρρυθμίσει που απαιτούνται. Τι θα περιμένατε από μια υποψήφια χώρα. Θα περιμένατε να γνωρίζει ότι για να μέλος κάτω μέσω Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν πρέπει μόνο να κάνει όσα επιτάσσουν τα 35 κεφάλαια, να αποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις που αντικατοπτίζονται στα 35 κεφάλαια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει κράτος μέλος. Πρέπει να μοιραστεί πλήρως τις αξίες μας, τις αξίες αυτού του οργανισμού, αυτών των οργανισμών. Αξιοπιστία από την πλευρά μας. Τι λέω δηλαδή. Αξιοπιστία. Πριν από δύο χρόνια αποφασίσαμε για τους κανόνες του παιχνιδιού για τη διαδικασία. Πώς θα κυλάει η διαδικασία. Να τηρήσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Να μην τους αλλάζουμε τους κανόνες. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός για να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουμε και θα είμαστε το σημείο αναφοράς για τις ε, τουρκικές μεταρρυθμίσεις. Όλοι αναφερόμαστε στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία. Θα πρέπει να υπάρχει και δέσμευση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να αφοσιωθεί στην προσπάθεια αυτή τη διαδικασία, υλοποίηση τη διαδικασία. Δεύτερο σχόλιο. Αυτό το θετικό πρόγραμμα, η θετική ατζέντα που συζητήσαμε πέρυσι. Δούλεψε, έδωσε αποτελέσματα. Το λέω αυτό διότι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξάλληψε αυτή την οτροπία του εμείς το αξίζουμε. Κάτι που έχω ακούσει πολλές φορές από πολλούς Τούρκους εταίρους να το λένε αυτό. Το αξίζουμε να γίνουμε μέλη. Αναφέρθηκα και θετικά στοιχεία. Τα ανέφερε η Υπουργός, εκπρόσωπος της Προεδρίας, τα θετικά στοιχεία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι τα σημεία που βρήκαμε και αναφέραμε να τα συνδέσουμε για να δημιουργήσουμε ορμή, όθηση στην προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις να επιστρέψουν στη σωστή τροχιά και αυτή η διαδικασία να γίνει βιώσιμη. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός για να πλησιάσει η Τουρκία την Ευρώπη. Που καθορίζεται η Ευρώπη από το κάτω δικαίου, αξίες της, δημοκρατία και θεμελιώδης ε, ελευθερίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε και έτσι ολοκληρώνεται εδώ αυτό το σημείο στην εξέτασή του στην ημερήσια διάταξη με την παρέμβαση εξ του Συμβουλίου της κυρίας Κρέιτον. Έχετε τον λόγο κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους Ευρωβουλευτές για αυτό που πιστεύω ότι ήταν μια ευρύτερη συζήτηση, ευρύτατη συζήτηση. Καταδεικνύει αυτό σαφώς, σε μένα τουλάχιστον, ότι οι διαπραγματεύσεις αποκτούν μια νέα πρόθεση και ορμή αυτή τη στιγμή και συνεχίζονται να ενθαρρύνονται, συνεχίζονται να ενθαρρύνονται οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία. Αυτή είναι η καλύτερη πορεία προς το μέλλον και θα ακολουθήσουμε και αυτή την πορεία στο μέλλον, ενθαρρύνοντας αυθεντικές πραγματικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία εξέθεσα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις τους πολλούς τομείς όπου υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις σε σχέση με την Τουρκία. Δεν προτίθεμαι να επαναλάβω αυτή την απαρίθμηση αυτών των τομέων. Πιστεύω ότι απηχήθηκαν από αρκετούς ευρωβουλευτές αυτές οι απόψεις. Επίσης ε, υπογραμμίστηκε και στο ψήφισμα και όλες οι πλευρές έχουν να κερδίσουν από αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και της περαιτέρω ε, συνέχισης πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία. Από πλευρά μας η Προεδρία, από κοινού με τα κράτη-μέλη και από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράττουμε ότι είναι στο χέρι μας για να σημειωθεί πρόοδος. Και αυτό υπό την Ιρλανδική Προεδρία πρέπει να πω ότι ήταν κάτι σημαντικό και ελπίζω ότι θα σημειωθεί πρόοδος και κατά τα τέλη της Προεδρίας μας, περαιτέρω πρόοδος. Θέλω να ολοκληρώσω υπενθυμίζοντας ότι στο τέλος τέλος είναι η ίδια η βούληση και το στένος της Τουρκίας να προχωρήσει προς τα εμπρός που θα καθορίσει τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων. Έτσι λοιπόν το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο της Τουρκίας. Η πρόοδος της Τουρκίας να ανταποκριθεί στους όρους και ε, προϋποθέσεις στους γνώμονες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ο πρώτος και κύριος καθοριστικός παράγοντας πρόοδο στι διαπραγματεύσει δεν θα απαιτεί μόνο περαιτέρω προσπάθειε για περαιτέρω μεταρρυθμίσει, αλλά και ένα μεγάλο βαθμό πολιτικού θάρρου και πνεύματο ηγεσία από πλευρά τη τουρκική κυβέρνηση. Από πλευρά μα παρέχουμε την υποστήριξή μα προ περαιτέρω τέτοιε προόδου. Θέλω τέλο να τονίσω τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την πολιτική διεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμπλέκοντα του πολίτε, τα κράτη-μέλη έναντι της Τουρκίας σε δημοκρατικές διαβουλεύσεις και συζητήσεις. Κέρια σημασία ε, για την συνέχιση αυτής της σημαντικής ε, διαδικασίας για το μέλλον. Αξίζει να το επαναλάβουμε και να το επαναλαμβάνουμε αυτό επανειλημμένα. Θέλω να ευχαριστήσω τους Ευρωβουλευτές για μια καρποφοραγόνιμη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα την εισηγήτρια. Ευχαριστώ όλους. Γεια. σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Και με αυτή την παρέμβαση ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο. Έχουμε μια πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Προέρχεται από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η ψήφιση θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30 το πρωί. Αλλά δεν θέλω να εγκαταλείψουμε αυτό το σημείο χωρίς να συγχαρώ την κυρία Όμεν Ρόιτερ ως εισηγήτρια για αυτό το οποίο καταδείχθηκε με εξαιρετική συμμετοχή στη συζήτηση, με εξαιρετική